It's the same, like, I suppose you have the same problem. A ver, buenos días a todos. Con 10 minutos de... Καλημέρα σας. Με μία δεκάλεπτη καθυστέρηση θα αρχίσουμε και περιμένω μέχρι ότου λάβετε θέσεις όλοι. Πρώτο σημείο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να δεχτούμε τις Αλλαγέ στι τελευταίε στιγμές που έγιναν και που εμφανίζονται μόνο στην αγγλική διορθωμένη εκδοχή, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη ανακοίνωση, γι' αυτό θα σα πρότεινα να περάσουμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη, που είναι οι εφαρμοστέοι κανόνε στην εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, αλληλευτικών προϊόντων, δίθυρων ε, μαλακίων, εχινόδερμων κτλ. και των παραγόγων προϊόντων, προϊόντων τους από τη Γρυλανδία. Για να δούμε αν το βρω το θέμα στο φάκελό μου. Όπως θα θυμάστε, πρόκειται για μία πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ και όχι της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Είχαν ζητήσει την ε, γνώμη μας τον περασμένο Απρίλιο ήδη η νομική βάση που ήταν το άρθρο 213 της συνθήκης αφορούσε μια διαδικασία διαβούλευσης και όχι την νομοθετική διαδικασία της συναπόφασης. Εμείς με την ανεκτήμητη υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώσαμε ότι η η νομική βάση, το άρθρο 203 της συνθήκης δηλαδή, ήταν α, ακατάλληλη και κανονικά θα έπρεπε να επιλεγεί η νομική βάση για την κανονική νομοθετική διαδικασία. Βέβαια τότε είχαμε μια σειρά προβλημάτων εξαιτία και των σχεδίων διαχείρισης και θεωρήσαμε ως το θέμα, το θέμα αυτό ήταν ίσονο σημασίας, δευτερεύον. Γι' αυτό δεχθήκαμε αρχικά την διαδικασία διαβούλευση, παρόλο που είχαμε αναγνωρίσει την ακαταλληλότητά τη. Σκεφτήκαμε ότι μου θα ήταν εκείνη τη στιγμή να συσπηρωθούμε και να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας ε, για άλλα θέματα που ήταν προτεραιότητα για τότε και ήταν ε, τα σχέδια διαχείρισης. Μια και πρόκειται να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή, όσο μάλλον λαμβάναμε την ε, έκθεση αυτή. Ακούσαμε ότι το Συμβούλιο δέχτηκε την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε ε, κληθήκαμε και εμείς να επανεξετάσουμε το θέμα. Τότε είχαμε ζητήσει την γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε μια γνωμοδότηση που έχετε λάβει τους φακέλους σας και φαντάζομαι την έχετε διαβάσει, δικαίωσε το το Κοινοβούλιο, δηλαδή εμάς, την Αλληλευτική Επιτροπή, ως προς την πρόταση νομικής βάσης. Και μάλιστα το θέμα στηρίζεται στο πρωτόκολλο 34 του ειδικού καθεστώτος που εφαρμόζεται για τη Γρυλανδία. Το πρωτόκολλο 34, που απαρτίζεται από ένα και μόνο άρθρο, προβλέπει σαφέστατα ότι για τα θέματα εισαγωγής αλληλευτικών προϊόντων θα πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 43. Και το 43 για την ακρίβεια, όχι το 43.3 που αφορούσε το ΤΑΚ και ποσοστώσεις. Και μάλιστα και το άρθρο 204. Αποφασίσαμε λοιπόν, εγώ ειδικά που ανέλαβα την έκθεση ως πρόεδρος, να τροποποιήσουμε την έκθεσή μας μετά τις συστάσεις της γνωμοδότησης της Νομικής Επιτροπής και να υποβάλουμε προτάσεις με βάση τη νέα νομική βάση. Δεχόμαστε λοιπόν την ε, διτή νομοθετική διαδικασία της συναπόφασης με βάση τα άρθρα 43.2 και 204 της συνθήκης και από αυτή την άποψη θα σας παρουσιάσω την έκθεσή μου με τη νομική βάση που σας ανέφερα. Βέβαια, είναι περιττό να σας πω ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφωνούν με τη θέση μας, αλλά ήταν αναμενόμενο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν εσείς συμφωνείτε με την θέση για την νέα νομική βάση. Γι' αυτό και θα σας δώσω το λόγο. Πρώτα σε εσά, στα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής και μετά στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ. Θέλει κανείς το λόγο. Όχι, οπότε ας ακούσουμε τον κύριο Μάγερ από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σημειώνω τη γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Δεν είμαι εγώ νομικός εμπειρογνώμονας, αλλά για μένα είναι σημαντικό να γνωρίζω ότι τα μέτρα αυτά υποστηρίζονται από όλα από όλα τα συμβαλόμενα μέρη εφόσον αφορά τη Γρυλανδία και πρέπει να ε, υποστηρίξουμε από κοινού κάτι όλοι μαζί. Δεδομένου ότι θα γίνει νομοθετική πράξη για την ε, κοινή αγορά με τη Γρυλανδία σε αλλιευτικά προϊόντα. Ε, χαίρομαι που λύθηκε το θέμα της νομικής βάσης. Πιστεύω ότι είναι τυπικό θέμα, αλλά χαίρομαι που δεν υπάρχει καμία ε, αφισβήτηση πια της ουσίας. Σέβομαι τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι θα λυθεί αυτό, ότι μετά τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν πιστεύει ότι η σωστή βάση είναι το άρθρο 1. Μιλάμε για υγειονομικά μέτρα, είναι μέτρα που αφορούν τον τομέα της υγείας και εμείς έχουμε τη γνώμη ε, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ε, ενταχθούν στα μέτρα υγειονομικών ελέγχων των ε, προϊόντων αυτών, των ελευτικών προϊόντων. Γι' αυτό εμείς υποστηρίξαμε αρχικά το άρθρο 9 ως νομική βάση, αλλά ε, πιστεύω ότι μετά την γνωμοδότηση αυτή το θέμα ε, λύθηκε και ότι δεν θα υπάρχει πλέον ε, αμφισβήτηση της νομικής βάσης η οποία υπήρχε αρχικά. Είχαμε μια άλλη νομική βάση εμείς. Η ανακύκλωση του άρθρου 204 και του πρωτοκόλου 34 πιστεύω ότι αποκλείει το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε δηλαδή και τα δύο να το χρησιμοποιήσουμε γιατί το ένα ακυρώνει το άλλο. Το 204 ακυρώνει το 34 πρωτόκολλο και αντίστροφα. Δίνω το λόγο στον αδελφό μου. Δεν ξέρω εάν χρειάζεται να σας αναλύσω τη νομική θέση της Κομισιόν ή πιστεύετε ότι είναι σαφές το θέμα. Um, uh, Εμείς ε, από πλευράς Κομισιόν πιστεύουμε ότι το 198 μέχρι 204 άστρα της ε, συνθήκης ε, περιγράφουν ε, τα, τον, την νομική βάση για τα αλλιεύματα ε, περιλαμβανομένης και της Γρυλανδίας. Και ε, επίσης καλύπτουν τις μονομερείς σχέσεις με τα, τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν ένα ειδικό καθεστώς και δεν είναι ξεχωριστά κράτη-μέλη ή κράτη, τρίτα, τρίτα κράτη. Ε, περιγράφει, λοιπόν, το, περιγράφουν λοιπόν τα άρθρα αυτό τις ειδικέ σχέσεις ε, με τα OCT και δι της Γρυλανδίας και κάνουμε την παραχώρηση αυτή για μία εξαίρεση από τους τελωνιακούς δασμούς. Και ότι το θέμα αυτό καλύπτει ε, ε, υγειονομικούς κανονισμούς και δεν καλύπτεται από το πρωτόκολλο. Θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του, του πλαισίου συμφωνίας με τις περιοχές αυτές και να καλύπτεται από το 203 άρθρο και να μην καλύπτεται από το πρωτόκολλο. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να εφαρμόζουμε και τα δύο πράγματα. Και το γενικό πλαίσιο συμφωνίας και το, ε, άρθρο, και το πρωτόκολλο 34. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κατάλληλη βάση είναι το 203. Το άρθρο 203 της συνθήκης. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελε να δώσει μια απάντηση, δεν χρειάζεται. Δεν είστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε να απαντήσετε, είναι ευκαιρία. Κύριε Στέλλα, ε, yes, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να απαντήσω σύντομα. Καταρχάς, αν δείτε το σχέδιο πρότασης, και εξετάσετε το στόχο, το στόχο του ε, σχεδίου πρόταση ε, πρότασης, το άρθρο 3 λέει ότι αφορά τις εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφόρων προϊόντων και ότι οι εισαγωγές αυτές θα πρέπει να εμπίπτουν στις παρακάτω ε, ε, διατάξεις. Επανέρχομαι τώρα στην ε, Συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την νομική βάση τη Κομισιόν και, λέω ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα το 203 και το 204. Πιστεύω όμω ότι το 204 είναι το σωστό. Το 198 με 203 θα εφαρμόζεται για τη Γρυλανδία υπό ε, ειδικέ συνθήκες. Τώρα, τι λέει το πρωτόκολλο 34. Στο μόνο άρθρο, παράγραφος 2 του πρωτοκόλου, λέει όλα τα μέτρα τα οποία σχετίζονται με μέτρα εισαγωγής. Αφορά συγκεκριμένα τις εισαγωγές. Και το άρθρο 3 ε, της, ε, του σχεδίου πρότασης ακριβώς γι' αυτό μιλάει. Συνθήκες εισαγωγών, συνθήκες εισαγωγής των προϊόντων. Δεν βλέπω λοιπόν πώς μπορεί να καλυφθεί από αυτό το μοναδικό πρωτόκολλο άρθρο 2. Θα πρέπει πιστεύω να συναποφασιστεί το θέμα αυτό ώστε να μην υπάρχει αντίθεση, δικογνωμία και αντιφατική βάση. Πάντως, εμείς θα ακολουθήσουμε τη γνώμη της νομική υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της νομικής επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι μόνο η νομική υπηρεσία και η νομική επιτροπή στη γνωμοδότησή της είναι ξεκάθαρη και παρόλο που δεν είμαι εμπειρογνώμων σε νομικά θέματα με έχει πείσει απόλυτα η γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής και σας παροτρύνω να τη διαβάσετε κι εσείς. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μάγερ ότι επί τη ουσία δεν έχουμε πρόβλημα το πρόβλημα δημιουργείται με την ακολουθητέα διαδικασία και την νομική βάση. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε. Το Συμβούλιο είναι που είχε προβλήματα. Εμείς με την ουσία δεν έχουμε πρόβλημα. Με την ακολουθητέα διαδικασία έχουμε πρόβλημα. Μια ναι, και το Συμβούλιο άλλωστε μας έδωσε λαβή να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αποφασίσαμε να ξαναδώσουμε τη μάχη της νομικής βάσης. Έχετε το λόγο και πάλι κύριε Μάγερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να προσθέσω κάτι. Ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο που υιοθετήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου προσπάθησε να συγκεκριμενοποιήσει τον, το στόχο της πρότασης, το σκοπό. Άρθρο 3. Γενικοί κανόνες αφορούν τους υγειονομικούς ελέγχους μεταξύ της Ένωσης και της Γρυλανδίας Γι' αυτό τροποποιήθηκε λίγο για να καταστεί ο σκοπός ακόμα πιο ε, ξεκάθαρος, πιο σαφής. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε μετά την υιοθέτηση της ε, γνωμοδότησης. Καλώ, εμεί εμένουμε στη θέση μας. Η διορία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 4 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στη συνεδρίαση της 15ης. Οπότε ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξη και περνάμε στο σημείο 4 που είναι ο κανονισμός τεχνικών μέτρων με εισηγήτρια την κυρία Εστέλ Γκρελιέ. Το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, έμεινε εκρεμές μετά από το αίτημα πολλών ευρωβουλευτών να προβλέψουμε κάποιο χρόνο συζήτησης για τις τροπολογίες πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Εγώ είπα ότι από εδώ και πέρα οι εκθέσεις που συγκεντρώνουν πολλές τροπολογίες επί της ουσίας θα εξετάζονται πριν την ψηφοφορία στην Αλληλευτική Επιτροπή. Ως τούτου και στην περίπτωση αυτή δεν είχα κανένα πρόβλημα να δεχτώ το αίτημα των Ευρωβουλευτών, ε, κυρίως των συντακτών τροπολογιών, να προβλέψουμε χρόνο για συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γκρελιέ, και κατόπιν ε, θα αρχίσει η συζήτηση και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πένα, στον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής. Oui, Madame la, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου ε, που υπέβαλαν τροπολογίε επί συγκεκριμένη έκθεση. Πρόκειται για τροπολογίε που αφορούν κυρίω την ουσία του κανονισμού είτε για την αύξηση είτε για τη μείωση των ε, αλληλευτικών ικανοτήτων. Πρόκειται για μια, ε, ένα αίτημα παράταση, ένα αίτημα παράτασης για επιπλέον για μερικά χρόνια ακόμα, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 είναι κρίμα που πρόκειται για μια νέα παράταση, γιατί στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε συμφωνήσει για την έγκριση ενός νέου κανονισμού. Είχαμε πει λοιπόν 18 μήνες επιπλέον παράταση. Είναι σημαντικό το θέμα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για κοινωνικούς και για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ε, αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, γιατί αφορά και τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες του κλάδου και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και γι' αυτό ακριβώς τα τεχνικά μέτρα για μας χρήζουν ιδιαίτερης πιο ε, περιστατωμένης προσοχής ε, και στο πλαίσιο ολόκληρη αναθεώρηση του κανονισμού. Και γι' αυτό ακριβώ πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί μια απόφαση πιο μακροχρόνια. Και θα ήθελα γι' αυτό ακριβώ το λόγο να αναφερθώ στι τροπολογίε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ε, οι κατάλληλε. Είναι. Απλώς νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο συγκεκριμένες μελέτες ε, επιπτώσεων από αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή και πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε σε επιστημονικά στοιχεία. Νομίζω ότι η κατάσταση του επιτάσσει, ξέρω ότι το ε, συζητήσαμε και καλά κάναμε και το συζητήσαμε. θα έλεγα καλύτερα οι τροπολογίες ε, επί της ουσίας ε, να αναβληθούν καλύτερα μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευθεί να προβεί σε μελέτες ε, επιπτώσεων τις οποίες θα γνωστοποιούσε στους ευρωβουλευτές ε, και το λέω αυτό και στο πλαίσιο των τροπολογιών ε, αλλά και γιατί θα υπάρξουν και αξιολογήσεις γενικότερα τις οποίες έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του ζητήματος. Το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και για τις μελέτες και για τις αξιολογήσεις ε, γιατί ούτως ή άλλως και η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλεκτικής πολιτικής έχει τεθεί. Λοιπόν, Ελπίζω να, να βγω ζωντανή από την αίθουσα, ελπίζω να μην ε, δημιουργηθεί πρόβλημα με το αίτημά μου να μεταφέρουμε για κάποια στιγμή στο μέλλον ε, τις ε, τροπολογίες ουσίας, γιατί αν ψηφίσουμε σήμερα πρόχειρα και επιπόλαια θα μας ε, πούν ότι δεν λάβαμε υπόψη όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ε, ότι δεν ε, λάβαμε υπόψη όλες τις μελέτες, όλες τις αξιολογήσεις και δεν σημαίνει ότι η ψηφοφορία μας δεν θα είναι ουσιαστική, απλώς ότι δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τις τροπολογίες επί της ουσίας του κανονισμού. Αυτά ήθελα να σας πω σε σχέση με τα επιχειρήματα που ακούστηκαν για την συγκεκριμένη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω πρώτο το λόγο στους ευρωβουλευτές και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάσει τις τροπολογίες και τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω την κυρία Γκρελιέ για την εισαγωγή της. Αλλά, κυρία Γκρελιέ, μας είπατε ότι θα έπρεπε να ακούσουμε τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Οι τροπολογίες ε, έχουν προέλθει από τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Οι τροπολογίες συγκεκριμένα αφορούν ε, τον τομέα 7 που είναι η Δυτική Σκοτία και η θάλασσα της Ιρλανδίας. Οπότε το να ζητάτε να δείξουμε κάποια συμπαράσταση. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη, ήδη ε, ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες υπό, έντονες, υπό έντονους περιορισμούς. Μιλάμε για την αλληλεία στη Δυτική Σκοτία και στην Ιρλανδική θάλασσα. Και ένας από τους λόγους που έχουμε θέσει τις συγκεκριμένες τροπολογίες είναι ο εξής. Όταν ε, συμφωνήθηκαν αρχικά τα τεχνικά μέτρα ε, αφορούσαν σχέδια ανάκρισης του βακαλάου τα οποία αφορούσαν μία περίοδο 12 μηνών και αναμενόταν ότι αυτή η περίοδος των 12 μηνών θα ήταν επαρκής για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του βακαλάου. Και τώρα προσπαθούμε και πάλι να τα ε, ε, παρατείνουμε. Δηλαδή μιλάμε για μέτρα που ήταν κατεπήγοντα και αυτό που κάνουμε ε, τώρα είναι ζητούμε rollover χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς ζητούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και είναι αυτό το οποίο ακριβώς εσείς κυρία Γκρελιέ ζητάτε. Οπότε τα τεχνικά μέτρα δεν ε, ενδεχομένως να μην οδηγήσουν στην ανάκτηση των αλλιευμάτων ε, από τους αλλιείς ε, στην ε, Δυτική Σκοτία, οι οποίοι όλο και περισσότερο επιλεκτικοί πρέπει να είναι στα αλλιεύματά τους. Δηλαδή να υπάρχουν τα συγκεκριμένα μεγέθη δικτυών για ορισμένα ψάρια που αλληλεύονται στην περιοχή εκείνη ή για παράδειγμα μικρότερα αλλιευτικά σκάφη κάτω των 50 μέτρων για αλληλεία εκτός από το Βακαλάο ε, στην βορειοδυτική πλευρά της Σκωτίας. Μήπως θα μπορούσα να συνεχίσω και για τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ε, τροπολογία 5. Ε, ζητούμε μικρότερα ε, δίχτυα για το ε, εν λόγω αλίευμα γιατί έχουν ε, αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές και υπάρχει περίπτωση σε, ε, να, να καταρρεύσει ολόκληρη η αγορά. Είναι λοιπόν σημαντικό να ζητούμε για τη Ζαγκέτα συγκεκριμένα μείωση των ε, ε, δικτυών, των ματιών των δικτυών. Επίσης, ζητούμε συγκεκριμένα για το ψάρι κρόφης και για την περίοδο των καλοκαιρινών ε, ε, μηνών, να περιοριστεί σε, περίοδο, να περιοριστεί σε ε, ποσότητα ενός εκατομμυρίου τόνων. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλείς που ζουν από το συγκεκριμένο αλίευμα στην, στη βορειοδυτική σκοτία. Γιατί διαφορετικά καταστρέφονται τα αλίευματα. Όσον αφορά τροπολογία 9 προστασία των ε, σκαφών που αλλιεύουν καραβίδα γιατί ούτως ή άλλως τα παραλιεύματα δεν είναι μεγάλα σε εκείνη την περιοχή και η τροπολογία 10 αφορά τα σκάφη που είναι μικρότερα από 15 μέτρα στην βορειοδυτική ε, περιοχή της Σκοτίας που είναι και η περιοχή 7 γιατί ε, τα τεχνικά μέτρα που έχουν ε, επιβληθεί είναι πάρα πολύ αυστηρά και οι αλληλείς δεν μπορούν δεν έχουν τα σκάφη αυτά δεν αλιεύουν βακαλάο αλλά εισόδημα. εντελώς αδύνατο να μπορέσει κανείς να αλιεύσει ή αλλως τα σκάφη αυτά δεν αλλιεύουν βακαλάο, αλλά ο, οι κανονες που ισχύουν σημαίνει ότι είναι εντελως αδύνατο να μπορέσει κανεις να ε, μπορέσει να αλλιεύσει ζαγκέτα ή εγλεφίνο ή άλλα ψάρια. Υπάρχει επίσης και ένα πρόβλημα με τα σκάφη των κάτω των 15 μέτρων, ε, ζητήματα υγιεινής, ε, γιατί 80 χιλιόμετρα πηγαίνουν από το λιμάνι από το οποίο ξεκινούν και τα υποχρεώνουμε, αν συνεχίσουμε με τα τεχνικά αυτά μέτρα, να ε, πάνε ακόμη μακρύτερα και αυτό ε, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Η τροπολογία 11 θέλει να αποσαφηνίσει το μάτι το διτό που χρησιμοποιείται για το ψάρι μπόρφης ε, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ιρλανδούς αλληλείς, αλλά και για τους Σκο... Ε, Σκοτσέζους αλληλείς ε, και οι Υπουργοί αποφάσισαν να δώσουν τη δυνατότητα για 67% μέγιστο επιτρεόμενου αλλιεύματος για το είδος αυτό του ψαριού, το οποίο όμως αλλιεύεται με πολύ μικρότερο μάτι δικτύου από 32-44 χιλιοστά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μάτι δικτύου συγκεκριμένα για το αλλιεύμα του ψαριού ψαριού ε, Είναι λοιπόν ε, πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι τροπολογίες για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε τα τεχνικά μέτρα, να εξασφαλίσουμε το επάγγελμα της αλληλεία στις περιοχές αυτές, της Σκοτίας και της Ιρλανδίας και μιλάω επίσης κυρίως για τα σκάφη που είναι κάτω των 15 μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Στέλ για την ε, ε, δουλειά της ε, που είναι πολύ καλή όπως πάντα και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι συμφωνώ με την ανάλυση της. Είναι λίγο υπερβολική η θέση του συναδέλφου Στρούαν. Είναι πάρα πολύ ζωφερή η εικόνα που παρουσιάζει στο δικό του τομέα. Βρίσκω ότι είναι λίγο υπερβολικά όλα αυτά. Θα ήθελα να σα πω λοιπόν τη δική μου άποψη. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για όλον τον αλληλευτικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε είναι ο Ιρλανδικό, είτε είναι ο Ισπανικό, είτε είναι ο Ιταλικό. Ο σκοπό είναι η παράταση ενό προσωρινού καθιστώτο ε, τεχνικών μέτρων, ε, η οποία κατά τη γνώμη μου, αν δεν υπάρξει τροποποίηση, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει, να ε, αποφευχθεί ένα κενό νομικό μέχρι το 2013, κάτι το οποίο δεν θα ήταν καλό για την προστασία των αλλιευμάτων. Αν δηλαδή σήμερα τροποποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτός ε, από τον τύπο όπως ανέφερε η κυρία Γκρελιέ, υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει η διαδικασία, να αρχίσει πάλι μια εις συζήτηση και επί της ουσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης δυσκολεύουμε και τη ζωή των Ευρωπαίων αλλιέων. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα επί της ουσίας όπως είπε η κυρία Γκρελιέ. Άλλωστε έχει υποβάλει και εκείνη μια συγκεκριμένη τροπολογία από αυτού που αναφέρεται στη μορφή του κειμένου με την οποία συμφωνώ απολύτως. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμω ε, για την τροποποίηση των τεχνικών μέτρων σε συγκεκριμένε αλλιευτικέ ζώνε, όπω ε, είπε και ο κύριο Στίβενσον. Επίση, θα ήθελα να σα πω ότι περιμένουμε ακόμη μια μελέτη επιπτώσεων. Το είπε και η συγκήτρια προηγουμένω. Αυτή τη στιγμή τα τεχνικά μέτρα ε, πρέπει, να, πρέπει να περιμένουμε τα, την μελέτη αυτή επιπτώσεων για να δούμε τι θα κάνουμε με την παράταση όχι των τεχνικών μέτρων. Νομίζω λοιπόν ότι καλύτερο θα ήταν να ε, συζητήσουμε τα τεχνικά μέτρα τότε όταν θα υπάρχει η νομοθετική πρόταση, να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και να συζητήσουμε και για την ε, μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Γιατί νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ νωρί δεδομένων των γνώσεων που έχουμε να κάνουμε σοβαρές τροποποιήσεις όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα. Εγώ λοιπόν, ε, εκτό από τι τροπολογίε κυρία Γκρελίου, όλες οι υπόλοιπε θα τις απέριπτα ή εν πάση περιπτώσει θα μπορούσα να δεχτώ και την 4 και την 5 που δεν αφορούν την ουσία, αλλά σε γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να τροποποιηθεί αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Γκάλαχερ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και για την καλοσύνη που είχατε να συμπεριλάβετε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα για συζήτηση. Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια. Είναι θέμα συγκινησιακά φορτισμένο, κοινωνικό, αφορά τους, ε, τον κλάδο και όπως είπε ο και ο Στριόν Στίβενσον, είναι τεράστιες οι συνέπειες για τις μικρές εμβέλειες σε συγκεκριμένες ζώνες. Εγώ το 1994, πριν έρθω στο Κοινοβούλιο, ήμουν ένθερμο υποστηρικτή των τεχνικών μέτρων συντήρηση. Τα τεχνικά όμω μέτρα συντήρησης θα πρέπει να εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο και ουσιαστικά. Και τώρα ζητάμε rollover γιατί πραγματικά δεν έγιναν μελέτες επιπτώσεων. Είπαμε 18 μήνες, 12 μήνες αρχικά, μετά έγιναν 18, τώρα ζητάμε άλλους 18 μήνες παράταση ώστε όσους έδειξαν ανεύθυνη συμπεριφορά να διενεργήσουν τώρα τις μελέτες επιπτώσεων. Για να γίνουν μελέτες επιπτώσεων πρέπει κανείς να πάει επί τόπου και να διαπιστώσει πώς οι τροπολογίες μας θα επηρέαζαν την συνολική κατάσταση των αποθεμάτων. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν αμεληταίες οι συνέπειες. Και δεν μιλάμε για μεγάλα σκάφη, μιλάμε για μικρά αλλιευτικά σκάφη που δεν μπορούν πια να αλλιεύσουν στην ε, περιοχή αυτή. Θα πρέπει να πάνε 80 ε, μίλια ανοιχτά στον Ατλαντικό ή Νότια. Δεν έχουμε καμία συνείδηση να εξωθήσουν αυτούς τους ανθρώπους από τόσο μακριά για να μπορέσουν να κάνουν τις πληρωμές ενώ αν γίνουν δεκτέ οι τροπολογίε μα, θα μπορέσουν αυτοί οι να αλλιεύσουν εκεί, χωρί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα αποθέματα γάδου. Και νομίζω ότι μια τροπολογία για ειδικά αλλιευτικά εργαλεία, tangle nets, είναι πολύ σημαντική. Γιατί ουσιαστικά μόνο καραβίδες θα μπορούν να, να αλλιεύουν με τα ε, δίχτυα αυτά. Ούτε ζαγκέτες, ούτε πεσκαντρίτσες, ούτε ούτε άλλα ψάρια. Μιλάμε εδώ για πραγματικούς ανθρώπους, για ψαράδες που δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα. Με τις τροπολογίες μας δεν πρόκειται να έχουμε κανέναν ε, ριζοσπαστικό αντίκτυπο. Απλώς ε, θα βοηθήσουμε τους αλληλείς. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέγεθος για όλους. Μία λύση για όλους. Γιατί κάτι που ισχύει για ένα τμήμα της Ένωσης είναι κατάλληλο για άλλη περιοχή της Ένωσης. Και αυτό είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα όπου θα πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό. Και μαζί με τους ε, συντάκτες των τροπολογιών σας διαβεβαιώ ότι το σκεφτήκαμε από όλες τις πλευρές. Δεν είναι μια ισοπεδωτική ενιαία λύση η πανάκια για το πρόβλημά μας. Είναι και θέμα κοινού νου, κοινή λογική. Δεν είναι για πολιτικού λόγου που πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο και για τεχνικού λόγου. Γιατί όσοι τα πρότειναν αυτά αρχικά και κατέθεσαν τα μέτρα τεχνική συντήρηση, είτε ήταν παραπληροφορημένοι, είτε ανίδεοι ω προς τι συνέπειε όλων αυτών των μέτρων τεχνικής ε, υποστήριξη που υπέβαλαν. Και υπάρχει και ένα νέο σύστημα, Πρόεδρε, τώρα, που αν εξετάσουμε τις τροπολογίες θα φαινόταν ότι δεν τροποποιεί πλήρω το θέμα. Είναι λίγες λέξεις μόνο. Κοιτάξτε, αν κοιτάξετε είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά τις τροπολογίες, θα δείτε ότι προκύπτει ότι μόνο στην τροπολογία 7, η μόνη τροπολογία φορά τα tangled nets και το lesser spotted dog Πού είναι τα ε, dogfish, τα σκυλόψαρα, πού θα μπορούσε να μας ε, εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προσπαθούμε να κάνουμε και τι προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Είναι πραγματικά γελίο που δεν το συμπεριλάβαμε. Και έκθεση Hudson. Μιλάει για τα τάγκλινετς, για τη συμπερίληψη αυτή. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Κοίτα Επίσης για τα 120. Ποιος είναι αυτός ο, αυτή η διοφία που είπε 110 mm, ε, ε, χιλιοστά είναι το σωστό ε, μέγεθος για τα διάκαινα. Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει κάτι τέτοιο το, την αλία του εγλεφίνου. Παρακαλώ, δώστε μου μία ευκαιρία να εξηγήσω με απλά λόγια ότι το σημείο 11 δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα μέτρα τεχνικής συντήρησης ούτε τροποποιεί τον κανονισμό του 98 του Συμβουλίου. Ουσιαστικά, τον 850-98, ουσιαστικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα τάκια της ποσοστώσης του Δεκεμβρίου. Και στα συμπεράσματα και στη δήλωση αναφέρονται για το Borefish η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες στις αρχές του 2011 προκειμένου με βάση τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία να προβλέψει κατάλληλα διάκαινα ματιού για, τις, για την αλία του είδους μπόρφης και να προβλέψει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό. Το είδος αυτό, το Borfish, είναι ένα νέο πελαγικό αλλιευτικό είδος. Και ουσιαστικά σε αυτή την αλληλεία πρωτοστάτησε ο δανικός αλλιευτικός κλάδος, η, η, δανική αλληλεία. Αλλά και για τη Δανία και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τους υπόλοιπους ε, που αλλιεύουν αυτό το είδος είναι σημαντικό για όλους για όλες τις χώρες που διαθέτουν ε, το είδος αυτό και μιλάμε για 20 εκατομμύρια περίπου. Θέλουμε μια νομική βάση. Γιατί υπάρχουν ε, μεγέθη δικτυό για πολλά αλλιευτικά είδη και έχουμε και ένα συνολικό, μια συνολική διάταξη που λέει όλα τα υπόλοιπα είδη θα πρέπει να αλλιεύονται με, με δίχτυα που έχουν 100, ε, διάσταση 100 χιλιοστά διάκαινα. Πραγματικά δεν έχει νόημα αυτή η, πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε 32 με 54 χιλιοστά είναι το κατάλληλο διάκαινο. Με 100, 100 χιλιοστά τι να πρωτομείνει στο δίχτυ. Στις 15 Δεκεμβρίου είχαμε μια συνεδρίαση και ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τροπολογία και να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την έκθεση ως φορέα για να προωθήσουμε την απαιτούμενη νομοθετική ρυθμίση. Για το Συμβούλιο Επιτροπή ήδη είπαν ότι θα αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί να περιμένουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο μήνα του έτους αν μέχρι το Μάρτιο δεν ε, έχουμε μία πρόταση, μέχρι να εφαρμόσουμε τη διαδικασία της συναπόφασης θα περάσει πολύ καιρό. Έχουμε 32.000 τόνους, δεν υπάρχει πίεση για αυτά τα αλλιευτικά αποθέματα. Νομίζω είχε νόημα που δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με την κοινή αλληλευτική πολιτική του 1993, γιατί στηριχθήκαμε σε ιστορικές επιδόσεις. Είναι ευκαιρία τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, και τη Δανία που πρωτοστάτησαν σε αυτή την αλία που ούτως ή άλλως μετριάζει την πίεση για άλλα αλευτικά είδη. Γιατί να μην γίνει διαφοροποίηση μεταξύ αυτού του αλευτικού είδους και όλων των άλλων τεχνικών μέτρων. Χρησιμοποιούμε ως ευκαιρία και ως φορέα αυτή την έκθεση για να ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει πρόταση. Και έτσι είναι κλάβει αυτή την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή την, ε, το διάβημά μας. Δεν θέλουμε να μπούμε στα δικά της χωράφια, αλλά να τη βοηθήσουμε. Νομίζω ότι έτσι θα βοηθήσουμε και τους αλληλείς μας. Και σας θέρμο παρακαλώ. Μην εμείνετε στη θέση που ακούστηκε το Στρασβούργο. Κάντε μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτής της τροπολογία για το είδο Μόρφη και τι υπόλοιπε τροπολογίε. Είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε η έκθεση αυτή. Και μάλιστα μας είπαν το Δεκέμβριο ότι ήταν παράνομο. Λάθος. Και το... Ε, Μα δικαίωσε τελικά και η νομική υπηρεσία ότι ήταν απόλυτα νόμιμη και θεμητή αυτή η ενέργεια. Να δείξουμε στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε μια ρεαλιστική επιτροπή και ότι μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και σκεφτείτε το και εσείς λίγο μέχρι το απόγευμα. Εξετάστε την τροπολογία και θα δείτε ότι έχει νόημα. Πρόκειται για μια αλία που δεν, ε, δεν επηρεάζει καθόλου ε, ή δεν ασκεί καμία πίεση στο αλληλευτικό είδος. Γιατί λοιπόν να μην δεχτούμε αυτή την τροπολογία. Και για το 11, η τροπολογία 11 δεν είναι καθόλου μέτρο τεχνικής συντήρησης. Διαχωρίστε τις τροπολογίες. Μερικοί λένε ας αφήσουμε την συναπόφαση, άλλοι λένε να την ε, υποστηρίξουμε. Εμείς είχαμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα επιμείνουμε στην απόφαση, Συναπόφαση. Και το κάνουμε και για τη Χιλή. Και εγώ αντιτάχθηκα τότε στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ θα πρέπει να λυγίσουμε και να εμείνουμε στη δική μας θέση. Θα ήθελα να ζητήσω και από του επόμενου ομιλητέ να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια σχόλια και παρακαλώ να είστε και πιο λακωνικοί, γιατί έχουμε πολλέ ε, εκθέσει στην ημερήσια διάταξη και πολλού ε, ομιλητέ που ζήτησαν το λόγο. Κύριο Χαρτόν. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον κύριο Στίβενσον να αναλύει πολύ ε, ε, ενδελεχώς τα τεχνικά μέτρα και τους διάφορους λόγους και τα επιχειρήματα. Και συνήθως ε, μιλούσε για τις τροπολογίες αυτές και τη θέση της Σκοτίας, της Ιλλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς πρέπει να κοιτάμε ακριβώς γενικά τα μέτρα αυτά και να μην εγκρίνουμε μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν, δεν αποκρίνονται στον ε, αρχικό μας στόχο. Ε, δεν συμφωνώ ε, με το επιχείρημα ότι μέτρα που εφαρμόστηκαν για 12 μήνες ως επίγοντα πρέπει να ε, παραταθούν για άλλους 12 ή 18 μήνες και μετά να δοθεί πάλι παράταση για 18 μήνες. Όχι 18 μήνες από σήμερα, 18 μήνες παράταση από τον Ιούνιο ε, του 2012 όταν θα ε, ε, τελειώσει η προθεσμία. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για παράταση δύο ετών. Δεν συμφωνώ με αυτό. Η κυρία Γκριλιέ φαίνεται ότι επίσης από την Κομισιόν η αρχική περίοδος αυτών των μέτρων θα πρέπει να παραταθεί ε, για 18 μήνες γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ε, να εκδοθεί μία μελέτη επιπτώσεων. Μα τι στο καλό έκανε η Κομισιόν τόσο καιρό δεν εργαζόταν. Όχι, δεν εργαζόταν ε, και δεν μελέτησε τις επιπτώσεις τις οποίες δεν είχαμε προβλέψει, διότι υπήρχαν επιπτώσεις οι οποίες ήταν απρόβλεπτες απρόβλεπτες επιπτώσεις λοιπόν πρέπει να καταγράφονται και να μελετώνται ώστε να μπορούμε να ε, διαγράφουμε τα καινούργια μέτρα, ιδίως για την αλλήλεια μικρής κλίμακας. Θα πρέπει λοιπόν να, να τελειώσει και όλη αυτή η ιστορία των ε, απορρίψεων. Τι εννοώ τώρα με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Το ένα στοιχείο είναι η βιωσιμότητα. Ήδη ε, στο, στη Ζαγκέτα ε, δημιουργούνται προβλήματα λόγω της, ε, του χρησιμοποιούμενου μεγέθους ματιών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία απρόβλεπτη επίπτωση. Επίσης, τα όρια των ε, επιτρεπόμενων αλλιευμάτων έχουν πολύ δυσμενείς επιπτώσεις διότι αντί να μειώνουν αυξάνουν τις απορρίψεις. Αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε με τροπολογίες διότι ε, φαίνεται ότι αντί να καταργούμε ή να μειώνουμε το πρόβλημα ζητούμε, απαιτούμε περισσότερες απορρίψεις. Πράγμα παράλογο. Τώρα, νότιο-δυτικά της σκοτίες, τις περιοχές αυτές αλίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ε, πρόβλημα του μεγέθους ε, δικτυών για μικρότερα ή χαμηλότερα σκάφη, τετράγωνα μάτια, τα οποία, ε, τα οποία συνήθως αλλιεύουν νεφροπλοεία πόδα, τα οποία ε, όμως τα αλλιεύματα είναι ε, πολύ ε, χαμηλής ποιότητος και δεν πιάνονται από... Τα, τα αλλιεύματα τα οποία πιάνονται από αυτά τα τετράγωνα μάτια είναι πολύ, πολύ χαμηλής ποιότητος και διακυβεύουν την επιβίωση των ε, αλλιών στην νότιο-δυτική περιοχή της Σκοτίας. Δεν πρέπει λοιπόν σιωπηλά να δειχτούμε αυτό το πακέτο, ούτε, να μην υποβάλλουμε τροπολογίες ε, και να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ναι αυτό το πακέτο ε, είναι δυσμενές για τους αλείς, αυξάνει τις απορρίψεις, αλλά εμείς θα το περάσουμε σιωπηλά και χωρίς αντιρρήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό για την Επιτροπή μας, γι' αυτό ακριβώς έχω υποβάλει πιστεύω, πολύ ε, λογικές και ουσιαστικές τροπολογίες οι, οποία, οι οποίες δεν θα αλλάξουν το πνεύμα αυτή του κανονισμού, αλλά θα προσαρμόσουν την ουσία ε, στις ε, πραγματικές ανάγκες των αλλιέων αυτών των συγκεκριμένων περιοχών και επίσης δεν έχουν, ε, δεν έχουν ε, ε, αντιμετωπιστεί οι αντιρρήσεις που είχα από την πρώτη στιγμή που υποβλήθηκε αυτό το σχέδιο και με τα σχέδια της, της παρατηρήσεις, τα επιχειρήματα και τις αναλύσεις όσων έλαβαν το λόγο δεν, δεν με καθησύχασαν διόλου. Δεν καταλαβαίνω το, το σκεπτικό των επιχειρημάτων. Α, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουμε τους επιτόπου ε, παράγοντες και αλληλείς. Ήθελα να ρωτήσω, έχουν λάβει υπόψη τις, τα επιχειρήματα των φορέων και των αλλιέων από τη Σκωτία και την Ιρλανδία. Από ό,τι φαίνονται στις προτάσεις δεν έχουν λάβει υπόψη. Σας παρακαλώ και πάλι να είστε πιο σύντομοι στις παρεμβάσεις. Κύριε Πατράο Νέβες, σας ευχαριστώ. Εγώ υπέβαλα μία μόνο τροπολογία που δεν μπορεί να αποκλειστεί με μία μόνο κοντιλιά, μόνο με τα επιχειρήματα που μας παρουσίασε η συγγήτρια. Και εγώ συμφωνώ ότι οι τροπολογίες και οι θέσεις που υποστηρίζουμε εδώ θα πρέπει να έχουν μία επιστημονική θεμελίωση και τεκμηρίωση και να απορρέουν από τις επαφές μας με τους αλείς. Αυτά τα δύο κριτήρια όμως, το επιστημονικό και η ε, επαφή με τους ελείς, πληρούνται πλήρως στην τροπολογία μου που μιλά για άρση της απαγόρευσης μεταξύ 200 και 600 μέτρων των ε, αλληλευτικών εργαλείων. Και μάλιστα τον Οκτώβριο του 2010, πολύ πρόσφατα, απαγορεύθηκαν τέτοια δίχτυα μεταξύ 200 και 300 μέτρων, χωρίς να έχει ε, διενεργηθεί καμία μελέτη που να δικαιολογεί, να δικαιώνει, να συστήνει αυτή την απαγόρευση. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι άλλα παρελθόμενα δίκτυα χαίρουν ε, τέτοια ε, εξαίρεση. Παρόλο που στην περίπτωση αυτή δεν δικαιολογείται η απαγόρευση και που δεν ε, θεμελιώνεται από καμία επιστημονική μελέτη. Πρόκειται για ένα αλληλευτικό εργαλείο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αλληλεία πεσκαντρίτσας. Θα ε, πλήξει τα μάλα των τομέα και μάλιστα θα παροπλήσει ορισμένα αλληλευτικά σκάφη που είναι μικρής εμβέλειας αλίας. Δεν μιλάμε για μεγάλων διαστάσεων βιομηχανική αλία. Πρόκειται για έναν ήδη αποδυναμωμένο κλάδο και δεν μπορούμε να τον πλήττουμε περαιτέρω με τέτοιες απαγορεύσεις που ούτως ή άλλως δεν συνοδεύονται από επιστημονική επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση. Αναφέρεται ότι θα πληγούν εδώ οι καρχαρίες ή τα σκυλόψερα που θα εμπλακούν σε τέτοια δίχτυα. Αυτό δεν ισχύει. Είναι τελείως αναδαφικό. Και μάλιστα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το επιχείρημα. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό επιχείρημα, καμία επιστημονική μελέτη που να δικαιολογεί την απαγόρευση αυτών των δικτυών μεταξύ 200 και 300 μέτρων. Η απαγόρευση θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2010 και ήταν τελείως άκαμπτη η εφαρμογή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τελείως αδιάλεκτη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε καμία περίπτωση δεν ε, συνοδεύεται από επιστημονικά επιχειρήματα. Αν διατηρηθεί αυτή η απαγόρευση και αν σήμερα χάσουμε την ευκαιρία να επαναφέρουμε την κατάσταση σε αυτή που ήσχε πριν την θέσπιση της απαγόρευσης, που ούτως ή άλλως δεν δικαιολογείται επιστημονικά, αν δεν αποκαταστήσουμε την τάξη στην περίπτωση αυτή, θα χάσουμε την ευκαιρία να κρατήσουμε βιώσιμο βιώσιμο ένα κλάδο που ασχολείται κυρίως με την αλία της Πασκαντρίτσας και ουσιαστικά ε, στηρίζει ένα μεγάλο τμήμα της πορτογαλικής αλίας και επιπλέον θα δημιουργήσουμε μία ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία για το μέλλον. Γιατί στο μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να καταργήσουμε την απαγόρευση αυτή που, επαναλαμβάνω, αυθαίρετα θεσπίστηκε και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση τον Οκτώβριο. Είναι αδικαιολόγητη διατήρηση αυτής της απαγόρευσης και όσο επιτρέψουμε την παράτασή τη τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να αντιστρέψουμε αυτή την άδικη, αδικαιολόγητη και αθεμελίωτη επιστημονικά πρόταση. Νομίζω ότι είναι απόλυτα θεμητή η τροπολογία μου και ζητώ την υποστήριξη των συναδέλφων. Ο κύριος Καπόλα Σάντος, συμφωνείτε με την κυρία Πατράου, ελπίζω να μην μακρηγορήσετε τόσο πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με κάλυψε σχεδόν πλήρως η συνάδελφος και μάλιστα η τροπολογία μου είναι παρόμοια με τη δική της. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του κυρίου Καντέκ. Γιατί με την πρόταση αυτή δεν υποβάλλουμε καμία ε, τροπολογία. Και μάλιστα ε, αν ε, δεν υποβληθεί τροπολογία είναι το μόνο τεχνικό μέτρο που δεν παρατείνεται. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική θεμελίωση. Εμεί θέλουμε παράταση κατά μία διετία ενό μέτρου που ίσχυε μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε να προλάβουμε μέχρι, μέσα στην επόμενη διετία να συγκεντρώσουμε τα επιστημονικά πορίσματα. Γιατί τέτοιε επιστημονικέ πληροφορίε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Άλλωστε, η απαγόρευση αυτή επηρεάζει άμεσα 370 αλληλευτικά σκάφη, το 50%, το 50 από αυτά είναι ε, λιγότερο από 15 μέτρα και επηρεάζει και πλήττει 1.500 αλίες. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα επηρεαστούν και που βιο, αποκλειστικό βιοποριστικό τους μέσο είναι αυτή η αλληλεία και η απαγόρευση αυτή απολύτως αθεμελίωτη θα τους πλήξει άδικα. Θα ήθελα να στήσω την κατανόησή σας και την υποστήριξή σας για να περάσει αυτή η τροπολογία. Σας ευχαριστώ κυρία Χόντουστ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για την εργασία της και πάντοτε θεωρούσα ότι έχει κάνει έναν έντονο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, έναν εμπεριστατωμένο διάλογο με τους ενδιαφερόμενος του κλάδου. Από το 2013 είπαμε όλοι να ε, εμπεδώσουμε μια ευλογή, ε, ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική. Αυτό προϋποθέτει τη συμφωνία επί των στόχων. Να θέλουμε να ενδυναμώσουμε την αλληλεία, να την ε, αναπτύξουμε, να την προστατεύσουμε και στο τέλος της γραφής να έχουμε αρκετά ψάρια ώστε να μπορούν να κανοποιηθούν όλοι. Αυτό το οποίο συζητούμε τώρα δεν είναι μια νομοθετική πράξη, συζητούμε για έναν κανονισμό με την παράκληση της Κομισιόν για παράταση. Διότι η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτός ο κανονισμός δεν ε, επιτρέπει ακόμα μια ε, ολοκληρωμένη ανάλυση επιπτώσεων και μας είπε ότι ο κανονισμός, έχουμε ακούσει μεγάλες επικρίσεις ότι ο κανονισμός αυτός ε, τέθηκε ενισχύει χωρίς ε, μία ικανοποιητική νομική βάση. Αν πράγματι αυτό έχει γίνει, τότε θα πρέπει να δώσουμε ε, εύλογο χρόνο στην Κομισιόν να επεξεργαστεί εκ νέου αυτή την πρόταση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους μας για την κοινή αλλιευτική πολιτική Καταλαβαίνω, κατανοώ τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ε, όταν υπάρχουν προβλήματα στις ε, περιοχές τους και ε, αδυναμίες τις οποίες θέλουν να διορθώσουν και να καλύψουν. Κάνω όμως μια παράκληση να υποστηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν και σας παρακαλώ να μην βιαστούμε και να μην αποφασίσουμε εν θερμό διότι ε, όλοι θέλουμε να έχουμε μία σωστή νομική βάση και ε, μία απόλυτα στεγανή νομοθετική πράξη. Ε, δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε ότι αλλάξαμε κατεύθυνση και θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση, σας παρακαλώ, να αφήσουμε εύλογο χρόνο στην Κομισιόν, να μπορέσει να επεξεργαστεί το ζήτημα και να μην υπάρχουν δικογνωμίες. Παραδείγμα, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιφατικά συμφέροντα, ας πούμε, από πλευρά ε, σκιωδών εισηγητών και Κομισιόν ή της δικής μας Επιτροπής. Όμως, Ας μην, ας μην επικαλύψουμε τη νέα αλληλευτική πολιτική με την παλιά το 2013. Ας δώσουμε χρόνο στην Κομισιόν. Έχουμε και τον κύριο Ρωμέ Βαϊρουέδα και μια άλλη ομιλήτρια πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν, ομολογώ ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονα στα θέματα αυτά. Άκουσα τους συναδέλφους και διαπιστώνω ότι υπάρχει εδώ και μια εδαφική διάσταση ή θέμα εγκύτητες με πολύ σημαντικές κοινότητες αλήφτικες. Έμαθα όμως ε, κάποια στοιχεία για το ζήτημα αυτό και τα στοιχεία που συγκέντρωσα εγώ είναι κάπως διαφορετικά από αυτά που άκουσα εδώ στη συνεδρίαση. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση όπου στο Κάτεγα, Καλ Μάρθελ, στην Δυτική Σκοτία, στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Μιλάμε για ελευτικούς πληθυσμούς που βρίσκονται στα όρια της ε, εξαφάνισης, στα, στα όρια των αποθεμάτων. Οπότε, οφείλουμε να ομολογήσουμε την αποτυχία των ε, σχεδίων συντήρησης, γιατί δεν εξασφαλίζουν ε, ούτε διατήρηση, ούτε πολλαπλασιασμό αύξηση των αποθεμάτων. Είναι τραγική κατάσταση των αποθεμάτων. Και αν δεν γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και αναμενόμενες βελτιώσεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με πολιτικές που όπως ε, φαίνεται έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. Κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι η διαπίστωση ότι πολλές τροπολογίες ουσιαστικά προέρχονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μέλων. Το είδαμε και στην ε, συζήτηση από το Συμβούλιο με εξαίρεση δύο τροπολογίε που καταθέσαν οι υπόλοιπε τροπολογίε είναι, είναι ουσιαστικά τροπολογίε που κατέθεσαν οι κυβερνήσει στο Συμβούλιο. Οπότε έχουμε εδώ τη μάχη μερικών χωρών μεταξύ τους σε κάποια αποθέματα που ούτω ή άλλως βρίσκονται σε αποδυναμωμένη κατάσταση ή είναι ανεπαρκή. Οι πράσινοι έχουν καταθέσει δύο τροπολογίε αφέστατε. Στην πρώτη αναγνωρίζουμε την αποτυχία των σχεδίων αποκατάστασης και την ανάγκη να ληφθούν νέα μέτρα. Μπορεί να θεωρηθεί ριζοσπαστικό, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιοδήποτε σχέδιο συντήρησης. Επίσης, θα πρέπει να μειώσουμε τις απορρίψεις με ένα μέτρο και κυρίως με την εισαγωγή συγκεκριμένων περιόδων παύσης αλίας για να προστατεύσουμε τις ε, δύσκολες, ε, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναπαραγωγής, τα ευαίσθητα αποθέματα. Μπορεί να κρίνεται απαραίτητη παράταση του ισχύοντος σχεδίου συντήρησης ή αποκατάστασης, αλλά είναι ανεπαρκής. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε η έλλειψη επιστημονικής μελέτης. Οι περισσότερες τροπολογίες ε, στο Συμβούλιο απορρίφθηκαν από τη ΣΤΕΛΦ, γιατί ακριβώς κρίθηκαν ως ανεπαρκείς. Εμείς, ως Αλληλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχουμε, υιοθετήσουμε μια πιο υπεύθυνη στάση, να δείξουμε ότι συνειδητοποιούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο κύριος Γκάλαχερ και άλλοι μίλησαν για την κατάσταση του ελευτικού πληθυσμού. Αλλά αν εξαντληθούν τα αποθέματα, δεν θα έχουν αντικείμενο πια οι αιλείς. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι εξαιρετικά λακωνική. Για την έκθεση αυτή δεν υπάρχει ούτε επιστημονική βάση, ούτε μελέτες επιπτώσεων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν ποια θα είναι η ακολουθητέα πορεία. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Μίλησε για τροπολογίε ε, τύπου και για τροπολογίε ουσία. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαφοροποίηση, γιατί εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιε είναι οι τροπολογίε τύπου και ποιε είναι οι τροπολογίε ουσία. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις ερωτήσει και να υποβάλει και τα σχόλιά τη. Ο κύριο Πένα. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τροπολογίε αυτέ συνοψίζεται σε δύο αρχέ. Η πρώτη αρχή αναφέρθηκε και από κάποιου παρεμβαίνοντε είναι ότι ο κανονισμό μας είναι ένα κανονισμό που στόχο έχει να εξασφαλίσει τη συνέχιση ε, κάποιων μεταβατικών τεχνικών μέτρων που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση στόχος του κανονισμού δεν είναι η νέα συζήτηση για τα τεχνικά μέτρα. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι στις 30 Ιουνίου θα είμαστε σε θέση να παρατείνουμε τα τεχνικά αυτά μέτρα που είχαν εγκριθεί τότε από το Συμβούλιο. Τώρα, αν μας ρωτάτε ποιες τροπολογίες θα στηρίξουμε, η θέση μας επί της αρχής είναι όσο το δυνατό λιγότερες γίνεται. Γιατί όσο περισσότερες τροπολογίες έχουμε επιτάπητος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να καταλήξουμε στη συμφωνία για αυτές πριν τις 30 Ιουνίου και άρα τόσο πιο δύσκολο θα είναι να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια των τεχνικών μέτρων που είχε τότε εγκρίνει το Συμβούλιο και που κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέτρα σημαντικά για τη συντήρηση των αποθεμάτων. Όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ανέκαθεν τη θέση ότι οποιαδήποτε ουσιαστική τροπολογία των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να συνοδευτεί από μια ε, ανάλυση των οικονομικών και επιστημονικών επιπτώσεων τη από την Οικονομική και Επιστημονική Επιτροπή Ελίας. Όπω ξέρετε, οι περισσότερε από τι τροπολογίε αυτέ, είτε δεν ε, εξετάστηκαν από την Οικονομική Επιστημονική Επιτροπή Επιτροπή Ελίας ή ακόμη και αν εξετάστηκε σε ορισμένε περιπτώσει, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή άλλα τεκμήρια που να δικαιολογούν αυτέ τι τροπολογίε. Κρίνουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια προηγούμενη αξιολόγηση. Κάτι που δεν ε, έγινε από τη ΣΤΕΛΦ ή ακόμη και αν έγινε δεν ήταν θετικό το αποτέλεσμά της. Με μία εξαίρεση. Και θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Η μόνη ίσως τροπολογία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις είναι η τροπολογία 11 για το Μπόρφι, το βασιλάκι όπως ξέρετε θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Καταρχήν δεν πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή των τεχνικών μέτρων, απλώς για μια διευκρίνηση μίας ε, αφησημίας του κανονισμού 850 κάθετος 98. Ουσιαστικά γίνεται μια διευκρίνηση και όχι ουσιαστική αναθεώρηση του κανονισμού. Επίσης υπάρχει ε, έκθεση της Επιστημονικής ε, και Οικονομικής Επιτροπής Αλίας που τάσεται υπέρ της αποσαφήνισης του μεγέθους ματιών για την αλία του βασιλάκη, του Μπόρφης. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Γκάλεχερ, υπάρχει εγκεκριμένη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο που η Επιτροπή, Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να βρει λύση για το θέμα αυτό. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, όσο, το δυνατότερο, όσο λιγότερες αλλαγές τόσο το καλύτερο, Στόχο μα είναι να εξασφαλίσουμε την παράταση εφαρμογή των τεχνικών μέτρων και μετά την 30 Ιουνίου και εν ώψη της ανάγκης ανάλυση, τεχνικής ανάλυσης ε, των προτάσεων αυτών πριν την έγκρισή του. θεωρούμε ότι μόνο για μία υπάρχει θετική αξιολόγηση και τη τεχνική επιτροπή αλλά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την τροπολογία 11 για τον Μπόρφη, το βασιλάκι. Και κάτι άλλο, κυρία Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το θέμα που έθεξε η Συγγετρία κυρία Γκρελιέ σε ό,τι αφορά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, αξιολόγηση των τεχνικών μέτρων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συζήτηση για το σύνολο των τεχνικών μέτρων αποτέλεσε το αντικείμενο μιας πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάστηκε εδώ και στο Συμβούλιο το 2009. Όπως θα θυμάστε, η πρόταση αυτή απέτυχε. Όχι για τεχνικά θέματα, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη προαναγγείλει κάτι που είπαμε και στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση, ότι για τα τεχνικά μέτρα χρειαζόμαστε ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα, όπου θα έχουμε και περιφερειακές αποφάσεις, γιατί οι περιφέρειες είναι πολύ πιο κοντά στον ελευτικό κλάδο. Τότε, το 2009, αυτή η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο, γιατί εκλήθηκε ως απώλεια εξουσίας για το Συμβούλιο. Απέτυχε λοιπόν η πρόταση και αποσύρθηκε το 2010. Τώρα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε τώρα. Η Επίτροπος Δαμανάκη είχε πει στην Επιτροπή σας ε, ότι μία από τις ε, προτεραιότητε που έχει για την μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτική είναι η θέσπιση μια απλούστερης νομική βάσης για τη συναπόφαση που θα επιτρέπει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για μια πιο αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, στους αλείς και στα συστήματα συνδιαχείρισης κτλ. Με αυτή την προοπτική λοιπόν θεωρούμε ότι η επανεξέταση όλων των τεχνικών μέτρων απαιτεί νέα νομική βάση που ευελπιστούμε ότι το Δεκέμβριο του 2012 θα εγκρίνουν οι δύο πλευρές της ομοθετικής αρχής και εσείς, δηλαδή μαζί με το Συμβούλιο. Οπότε θα υιοθετηθεί ένα πιο αποκεντρωποιημένο, περιφερειοποιημένο σύστημα απόφασης και με αυτή τη ε, βάση θα υποβάλουμε μια καινοτόμα πρόταση τεχνικών μέτρων που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό 850 του 98. Τώρα, για να μην μας λέτε ότι αναβάλουμε παόριστον τη συζήτηση για τα τεχνικά μέτρα, σας διαβεβαιώνουμε ότι ήδη από τώρα θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τη νέα πρόταση, ώστε όταν εγκριθεί ο νέος κανονισμός που θα επιτρέπει την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, αμέσως μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει έτοιμη για κατάθεση την πρότασή της. Ήδη αρχίζουμε τις εργασίες έχοντα υπόψη αυτό το νέο πλαίσιο, ευελπιστώντα ότι οι συνομοθέτε θα υιοθετήσουν ένα νέο βασικό κανονισμό τη κοινή ελληνική πολιτική που θα επιτρέπει μια πιο αποκεντρωμένη λήψη των αποφάσεων. Αυτά κυρία Πρόεδρε, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα διέπει τις εργασίες μας για τα τεχνικά μέτρα. Και το επόμενο έτος, επόμενους 18 μήνες, θα ολοκληρώσουμε τις τεχνικές συζητήσεις, τις επαφές με τους ενδιαφερόμενους και την αξιολόγηση του νέου συστήματος για τα τεχνικά μέτρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω μόνο. Στην προηγούμενη διαδικασία που απέτυχε, είπατε η αποτυχία οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους, όντως, αλλά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν ήθελαν να αποποιηθούν ε, των εξουσιών τους και να τις εκχωρήσουν όλες στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ήταν λόγω της ε, προτινόμενης αποκέντρωση περιεφερειοποίησης, αλλά δεν θέλαμε να εκχωρήσουμε όλες μας τις εξουσίες, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητούσε όλες πια αποφάσεις να λαμβάνονται με τη διαδικασία ε, των Συμβουλευτικών Επιτροπών. Η κυρία Γκρελιά έχει το λόγο. Oui, non, moi Κοιτάξτε, εγώ ακούω διάφορα επιχειρήματα και συγκεκριμένα για την τροπολογία 11 για να μπορέσω να απαντήσω και στην προλαλή σα και να αναφερθώ και σε ορισμένα σημεία που θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να επανεξεταστούν. Τροπολογία 1 σημαίνει ότι πρέπει οι μελέτες επιπτώσεων να γίνουν. Ε, ε είχα πει ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν νομίζω ότι είναι καμία ε, πολύ σοβαρή προσθήκη. Τώρα, σε σχέση με τις τροπολογίες που τροποποιούν τα τεχνικά μέτρα και θα το ξαναπώ γιατί από ό,τι κατάλαβα εκλήφθηκαν αυτά που είπα κάπως διαφορετικά από, αυτό που το, ε, από αυτά που εννοούσα. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη και την άποψη του κλάδου, αλλά και την άποψη και τα επιστημονικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλουμε και την αξιολόγηση, επιστημονικά στοιχεία, ε, και αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Ο κάθε, ο κάθε ένας έχει τη δική του τοπική και περιφερειακή άποψη, όμως εδώ Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ προέρχομαι από περιοχή αλλιευτική και γνωρίζω πολύ καλά τι χρειάζονται οι αλληλείς και τι είναι τα τεχνικά μέτρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να τεθούν επιτάπητος όλα τα τεχνικά μέτρα για όλους τους στόλους και για όλες τις αλλιευτικές περιοχές. Δεν είναι δυνατόν ε, για λόγω, λόγω παράτασης ενός κανονισμού να δώσουμε κάποια, να ευνοήσουμε τη μία ή την άλλη ελευτική ζώνη, ε, περιμένοντας κάποια μεταγενέστερα τεχνικά μέτρα. Όχι, είμαστε εδώ βουλευτές για να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά, όχι να δούμε μόνο το Ιρλανδικό πρόβλημα ε, ή το πρόβλημα της, Σκοτίν, της Σκοτίας, γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε να συζητάμε ο καθένας το πρόβλημά του και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα βγούμε έχοντας συμφωνήσει από την αίθουσα πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, να μην δώσουμε μία πρόθεση σε αυτή την έκθεση που δεν ήταν η αρχική πρόθεση της έκθεσης. Ε, και το λέω αυτό ε, προσθέτοντας ε, ότι οι τροπολογίες πρέπει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι τροπολογίες ουσίας. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά όχι στο πλαίσιο της συγκεκριμένη έκθεσης και στο πλαίσιο του χρονικού ορίζοντα που είχε δοθεί στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Α μην αρχίσουμε τώρα αντιπαράθεση. Όλοι είχαν την ευκαιρία να εκφέρουν τη γνώμη του και τελικό λόγο τον έχει κανονικά η εισηγήτρια. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Αν έχετε ερώτηση, εντάξει, αλλά όχι να μας εκφωνήσετε πάλι ομιλία. Just a question. Μία ερώτηση μόνο προς την εισηγήτρια και την Κομισιόν. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών που ελέγχθησαν, που, που, λένε ότι ίσως να έχουμε μια περιφερειακή αντιμετώπιση σε μερικά χρόνια. Και αυτά που είπε η εισηγήτρια και η Κομισιόν, δηλαδή Εν τω μεταξύ θα, θα κολλήσουμε σε αυτόν τον κανονισμό που, που δεν είναι ικανοποιητικό, που δεν δουλεύει σωστά. Πώς το καλό θα εφαρμοστεί λοιπόν η προτινόμενη συντήρηση, τα μέτρα συντήρησης. Θέλετε να απαντήσετε εκ από Η κυρία Γκρελιέ. Εγώ νομίζω ότι απαντήσατε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο ρόλος της Επιτροπής, ο τρόπος ε, με τον οποίο θα, ε, ε, θα διαγράψουμε στο μέλλον την αλληλευτική πολιτική, αλλά δεν είναι ο στόχος συγκεκριμένης έκθεσης. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τα τεχνικά μέτρα περιμένοντας μια μεταγενέστερη εξέλιξη και αν υπάρξει περιφερειοποίηση, ο καθένας θα ψηφίσει, επιτροπολογία ή μη, αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχο τη συγκεκριμένη έκθεση είναι να παρουσιάσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Καταλαβαίνω το τοπικό πρίσμα, καταλαβαίνω την επιθυμία ε, που έχει ο καθένα να υποβάλει τροπολογίε προστατεύει τους δικούς του αλληλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε μια πιο ευρωπαϊκή συζήτηση προκειμένου. Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή στη συζήτηση και στην κυρία Γκρελιά, την εισηγητριά μα να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει το απόγευμα γύρω στις 5 μετά την ε, συζήτηση που θα έχουμε με την Επίτροπο Δαμανάκη. 5 με 5 και 10 να είστε παρόντες γιατί θα ψηφίσουμε την ε, έκθεση της κυρίας Γκρελιέ. Ολοκληρώσαμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 5 που προβλέπει την ε, συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη και το σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας. Υποφαινόμενη συγκίτρια για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να σας πω ότι οι Ομόσπονδες Πολιτείς Μικρονησίας είχαν με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρωτόκολλο, αλληλευτικό πρωτόκολλο. Πρόκειται για μια ιδιάζουσα χώρα γιατί απαρτίζεται από 607 νησιά είναι μια νησιωτική χώρα, βρίσκεται στο κέντρο του Ειρηνικού ωκεανού και όταν ε, σας μίλησα για την σχετική επιτροπή αλίας του Ειρηνικού πρόκειται για μια πλούσια αλληλευτική ζώνη που βρήθη των οειδών και ξηφία. Είναι 3 εκατομμύρια τα τετραγωνικά μέτρα, είναι η 13η ε, ως προς την έκταση αλληλευτική ζώνη του κόσμου. Είναι εντυπωσιακή η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μικρονησίας και οι στόλοι που αλλιεύουν κυρίως αυτή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μικρονησίας είναι η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ταϊβάν και η Κίνα. Και μάλιστα οι ομόσπονδες πολιτείες Μικρονησίας έχουν συνάψει και με τις χώρες αυτές αλληλευτικές συμφωνίες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προηγούμενο πρωτόκολλο που είχε διάρκεια τριετή προέβλεπε τις ίδιες αλληλευτικές δυνατότητες, 6 γρηγροί και 12 παραγαδιάρικα, 6.200 τόνους, ενώ 16.200 τόνους, τώρα έχουμε 8.000 τόνους. Η χρηματική αντιπαροχή ήταν ετησίως 559.000 ευρώ όπως προβλέπεται και στο ισχύον πρωτόκολλο. Οπότε η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοκόλων είναι ε, η χωρητικότητα αναφοράς που μειώθηκε στα, στους 600 τόνους. Είχαμε και κάτι παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προηγούμενο πρωτόκολλο πρότεινε την, την πρώτη δόση χρηματικής αντιπαροχής, την πρώτη ετήσια δόση και μάλιστα τέσσερα γρηγροί ζήτησαν άδεια και κατέθεσαν τα 15.000 ευρώ συν τους δασμούς και τους φόρους που έπρεπε να καταβάλουν. Μιλάμε για μια χώρα που απαρτίζεται από 607 νησί και βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Παρόλο που υπήρχε αίτημα τεσσάρων γρηγρή και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είχε προβλεφθεί στο πρωτόκολλο, ε, κατέθεσε την πρώτη δόση χρηματικής αντιπαροχής. Έχουμε διάφορα ανέκδοτα από την περίπτωση αυτή. Ε, ο λογαριασμό τη Μικρονησία δεν δεχόταν ευρώ, για παράδειγμα. Διάφορε τέτοιε ιστορίε, αδιανόητε, αλλά σε τέτοιε περιοχέ τόσο απομακρυσμένε μερικέ φορέ συμβαίνουν και αυτά, γι' αυτό και στην πράξη ποτέ δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο. Στα τέλη Ιανουαρίου τρέχοντο έτου, το Κογκρέσο των Ομόσπονδων Πολιτειών Μικρονησία θα κυρώσει αυτή την αλληλευτική συμφωνία. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασε αυτή η προθεσμία. Έγινε η κύρωση από το Κογκρέσο της Μικρονησίας. Γιατί με μια χώρα που έχει τόσα νησιά, πού να συγκεντρωθούν οι γερουσιαστέ. Γιατί μία φορά το χρόνο, δεν κάνω λάθο, συνεδρίαζαν οι γερουσιαστέ. Οπότε, αν περάσει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει να περιμένουμε του χρόνου για νέα κύρωση. Ερωτώ λοιπόν συνεδρίαση των τελών Ιανουαρίου ενέκρινε το Κογκρέσο των, ε, της Μικρονησίας στην ελληνική Ζώνη. Όπως ξέρετε η χώρα αυτή είναι μέλος της α, ε, Κεντροδυτικής ε, Αλληλευτικής Επιτροπής του Ειρηνικού. Σας είπα τις προάλλες τι συμβαίνει σε αυτή την περιφερειακή οργάνωση αλληλείας. Σας παραπέμπω στις πληροφορίες που σας είχα δώσει σε εκείνη την περίπτωση. Η χώρα αυτή συμμετέχει στη Συμφωνία Βιοπικιλότητα, Κλιματικών Αλλαγών, του Πρωτοκόλλου του Κιώτο κτλ. Αλλά μέχρι στιγμή δεν έχει κυρώσει καμία από αυτές τις συμφωνίες. Το νέο πρωτόκολλο, όπως σα είπα, ε, αντί για τριετή έχει πενταετή διάρκεια και φτάνει σε 8.000 τόνους από τις 16. Η χρηματική αντιπαροχή είναι η ίδια. η προκαταβολή που δόθηκε θα καταμεριστεί καταναλογία κατά αναλογία του επόμενου έτους, μειώνοντας αντίστοιχα τις τόσες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για τους εφοπλιστές που προέβησαν σε προκαταβολές. Κάτι άλλο που επισήμανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαίνεται ε, και στην έκθεση σε ό,τι φορά την πληρωμή των αδειών. Φυσικά θα πρέπει να γίνει η προκαταβολή ε, του ποσού άδεια. Αναφέρθηκε η πληρωμή των παρατηρωτών που θα πρέπει να συμμετέχουν στα γρηγρή. Ενώ τα παραγαδιάρικα δεν υποχρεούνται να φέρουν στο πλήρωμά τους και παρατηρητές. Γιατί ισχύει μόνο για τα γρηγρή η υποχρέωση αυτή. Αναφέρεται άλλωστε και η πληρωμή αυτή των παρατηρητών σε περίπτωση καταβολής του ποσού άδεια. Ενώ για τα παραγαδιάρικα δεν αναφέρεται τίποτα. Βέβαια εντάξει είναι δευτερεύον θέμα αλλά το αναφέρω και στην έκθεση. Στην έκθεσή μου λέω ότι το νέο πρωτόκολλο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ενισχύει και ε, κατοχυρώνει την απαραίτητη παρουσία του Ευρωπαϊκού Στόχου γιατί όπως είπα και τις προάλλες είναι αδιαφεσβήτητη και σημαντική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη της Μικρονησίας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας και να καταπολεμήσουμε τη λαθρέα παράνομη και άναρχη αλία. Επαναλαμβάνω, ο αληφτικός μας στόχος είναι ε, τέσσερα, έξι γρηγοροί και τέσσερα παραγαδιάρικα. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει περισσότερα σκάφη. Άλλωστε είμαστε η μόνη οργάνωση που κρατάει αμύωτη την δέσμευσή της και τη στράπτευσή της για την καταπολέμηση της ε, παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στοιχεία που δεν ε, επέτρεψαν την έμπρακτη εφαρμογή του πρωτοκόλου. Μιλάω για την ε, τακτική σύγκληση των μεικτών επιτροπών. Επίσης μιλάω για την post ε, έκθεση αξιολόγηση που είναι η μοναδική που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τελευταία που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να προβλέψουμε και μία αντιπροσωπεία για την περιοχή αυτή που είναι πολύ σημαντική είναι σημαντικό να έχουμε αντιπροσωπεία λοιπόν και για την περιοχή αυτή. Αυτό ζητάει και η post έκθεση αξιολόγηση και μάλιστα δικαιολογείται όχι μόνο με τις, από τι τρει αλληλευτικέ συμφωνίε ε, με τα νησιά Κυριμπάτη, Σολομόντα και τη Μικρονησία αλλά και γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια αναπτυξιακή στρατηγική στην περιοχή αυτή που, με σημαντικό κονδύλιο που, από το, που καταβάλλεται από το Αναπτυξιακό Ταμείο. Οπότε δικαιολογείται μεγαλύτερη παρουσία επιτόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, εκφράζω την ανησυχία μου για τα τεκτενόμενα στην ε, Κέντρο Δυτική Ελληνική Επιτροπή του Ειρηνικού και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει για καλύτερη συνειδητοποίηση και επαγρύπνηση των χώρων αυτών σε ό,τι αφορά τα συστήματα διαχείρισης, στήριξη των αποθεμάτων κτλ. Και η παρουσία μας επιτόπου θα βοηθήσει στην βελτίωση της κατάστασης κατά τη γνώμη μου. Ένα άλλο θέμα που θα το θίξουμε και επ' ευκαιρία των Σιχελών. Η σύνοψη της εξπόστα για τις Σεϊχέλες προβλέπει ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα αυτά και ιδιαίτερα σε σχέση με την αλληλευτική συμφωνία με τις Σεϊχέλες συνέβαλε ώστε η κυβέρνηση και η διοίκηση των Σεϊχελών να βελτιώσουν κατά πολύ την προσέγγιση τους ως προς την βιώσιμη αλία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλους ελευτικούς στόχους που αλλιεύουν, όπως είναι της Ταϊβάν, της Κίνας, της Κορέας, που σίγουρα δεν είναι και η πιο φανατική υπέρμαχη της ε, βιώσιμης η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη πιο σημαντική. Ο κύριος Στίβενσον με αντικατέστησε στην συνάντηση με τους βουλευτές της Μικρονησίας. Οι βουλευτές είχαν κάποιες αφιβολίες ως προς την σκοπιμότητα αυτής της αλληλευτικής συμφωνίας. Ξέρω ότι ένα τμήμα του πληθυσμού είναι κάπως δύσπιστο και απρόθυμο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ τη βιώσιμη αλληλεία, ενώ η Κίνα και άλλε χώρε δεν είναι τόσο ευαίσθητε προ το θέμα αυτό. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολα τα μέτρα ε, της Κίνας από ότι αυτά που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξού και η απροθυμία μερικέ φορέ του τοπικού πληθυσμού να συμμορφωθεί, να δεχτεί μια τέτοια αλληλευτική συμφωνία. Ελπίζω με το τωρινό πρωτόκολλο να μην επαναληφθούν τα προβλήματα ε, του παρελθόντος Τώρα, ω προς την πληρωμή, ελπίζω να γίνει στη Χαβάη, που είναι μία από τις ε, ομόσπονδες πολιτείες Μικρονησίας. Ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με την κατανομή της χρηματικής, καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας και για, όχι μόνο για τις αλληλευτικές δυνατότητες, γιατί τι να σου κάνουν τέσσερα γρηγροί και εννιά παραγαδιάρικα. Δεν μιλάμε τόσο για τη σημασία της αλίας, περισσότερο για την παρουσία μας που θα είναι μια εναλλακτική φωνή, μια φωνή που θα τάσεται υπέρ της βιώσιμης αλίας, υπέρ της, των συμφερόντων της αλίας και φυσικά κατά της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Το λόγο ζήτησαν ο κύριος Άντζες Πρεσέντο, ο κύριος Καντέκ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η κυρία Μπιλμπά, ο κύριος Πρεσέντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας. Θεωρώ ότι η συμφωνία με τις Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για τέσσερις πολιτείες που ουσιαστικά συμμετέχουν και στις, στις χώρες του Ειρηνικού. Είναι μία από τις οχτώ χώρες ε, του Ειρηνικού που το 2000 προσυπόγραψαν και τη Συμφωνία Κοτονού. Η Ελευτική συμφωνία αρχική προέβλεπε ένα ετή διάρκεια, οπότε θα έπρεπε να ισχύει από το 2007. Βέβαια με το πρώτο πρωτόκολλο δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τα ελευτικά δικαιώματα. Ελπίζουμε τώρα να εφαρμοστούν και εμπράκτως αυτά τα ελευτικά δικαιώματα. Αυτό που επισημάνατε κυρία κυρία Πρόεδρε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή τα δικαιώματα που καταβλήθηκαν, ε, η χρηματική αντιπαροχή που καταβλήθηκε στην πρώτη δόση αλλά που δεν ε, βρήκε αντίκρισμα στα δικαιώματα, ειδικά για τα τέσσερα γρηγροί που ε, κατέβαλαν τις πληρωμές, θα πρέπει να καταμεριστούν κατά αναλογία στο μέλλον. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που ανέκυψε και γιατί δεν μπορέσαμε να καρποθούμε αυτά τα δικαιώματα. Μήπως θα επαναληφθούν αυτά τα προβλήματα και στο δεύτερο πρωτόκολλο, γιατί οι στόχοι είναι ίδιοι. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αλληλευτικές δυνατότητες και απασχόληση, να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη αλληλεία, καλύτερη διαβούλευση θέματα αλίας, ασφάλεια νεφοδιασμού. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την ευαίσθητη ζώνη, προκειμένου να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη υπεύθυνη και βιώσιμης αλίας και στην πρόοδο της αντίστοιχη περιφερειακής οργάνωσης. Από αυτήν την άποψη είναι πολύ θετική έκθεση και θα θέλουμε να ακούσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα επιφέρει το νέο πρωτόκολλο. Τι θα αλλάξει το νέο πρωτόκολλο στην κατάσταση και πώς θα βελτιώσει τις αλληλευτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καντέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε και για την έκθεση. Μας εξηγήσατε πώς λειτουργούσε η Επιτροπή του Δυτικού Ειρηνικού, λίγο περίεργα, και ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απαραίτητη. Τώρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκθεση, για την αξιολόγηση εκ των υστέρων της Συμφωνίας 2007, το είπατε κι εσείς, μαθαίνουμε ότι τα πρώτα τρία χρόνια δεν, έχει κανένα στόχο, δεν, δεν έγινε κανένα στόχος του πρωτοκόλλου του στα πρώτα τρία χρόνια. Το είπε και ο συνάδελφο ε, Σάντσε ε, Πρεσέντο. Κανένα από τα ε, γρηγροί δεν αλλιεύσαν στην περιοχή. Δεν υπήρξαν αλλιεύματα από την περιοχή, ενώ η οικονομική συνεισφορά είχε καταβληθεί και είναι και αρκετά σημαντική. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε ποιο βαθμό είναι ενδιαφέρουσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένη συμφωνία και τι εγγυήσει έχουμε για το μέλλον για τα δικά μα αλλιευτικά σκάφη που έχουν ζητήσει άδειε αλλιεύση στην περιοχή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μόνο για την ε, καταπολέμηση τη παράνομη αλληλείας που θέλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα να επιμείνει στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί είναι προφανώ ε, εθνικό σπόρο η παράνομη αλληλεία στην περιοχή. Και επίση η Μικρονησία. Εκείνη ήδη ε, ζητά επιπλέον πράγματα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάντως επέμεινα στην ανάγκη υποστήριξη βιώσιμης αλίας και πάταξης της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλίας. Πρόκειται για μια ζώνη και μια περιοχή στην οποία ισχύουν πολλές αλληλευτικές συμφωνίες. Και είναι σημαντικό η ζώνη να χαρακτηρίζεται από συνθήκες για βιώσιμη αλία. επέμενα στο θέμα αυτό, γιατί με απασχολούσε ιδιαίτερα η εμπειρία που είχα από την ε, Αλληλευτική Επιτροπή του Κεντροδυτικού Ειρηνικού. Γι' αυτό επέμενα σε αυτό. Κύριε Μπιλμπάου, και εγώ είμαι υπέρ της ε, ανανέωσης αυτής της Αλληλευτικής Συμφωνίας. Όπως είπατε, η παρουσία του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Στόλου δεν είναι πολύ σημαντική, αλλά συμβολικά είναι απαραίτητη. Όντως, ε, η εμπειρία σας από την Λευτική Επιτροπή του Ειρηνικού που μας εκθέσετε την περασμένη εβδομάδα μας προβλημάτισε και μας ανησύχησε, γιατί είναι σημαντικό να εμείνουμε στη δέσμευσή μας υπέρ της βιώσιμης αλληλείας και κρίμα που δεν συμμερίζονται και άλλες χώρες ε, τις δικές μας ανησυχίες. Φυσικά θα, καλό θα ήταν να επεκτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές και στη ζώνη αυτή και συμφωνώ με την ανάγκη ε, της παρουσίας μας στη Μικτή Επιτροπή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και για την ε, σύσταση της αντιπροσωπείας, γιατί έχουμε συμφωνίες και με τους νήσους Σολομώντα, Κυριπάτη και με τη Μικρονησία, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε και αντιπροσωπεία και το είχαμε πει και σε όλες τις συνεδριάσεις. Θα πρέπει τα μέλη της Αλληλευτικής Επιτροπής ε, να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στην τεκμηρίωση που κυκλοφορεί και στα έγγραφα. Εξακολουθούμε να ζητούμε αυτή τη διαφάνεια. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλούμε για παράνομη αλία, διαπιστώσαμε σε διάφορες πρωτοβουλίες ότι συνδέουμε την παράνομη αλία με, με τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Αλλά ο Ευρωπαϊκός Στόλος εξασφαλίσει κάποια χέγγια και διενεργεί ελέγχους. Εμείς ε, ασκούμε με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο την αλία. Για τις αλληλευτικές αυτές συμφωνίες σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσει μια εκστρατεία ενημέρωσης, προβολής, ε, μεγαλύτερης δημοσιότητας για να αποδείξει ότι ο Ευρωπαϊκός Αλληλευτικός Στόλος, όπου και να λιεύει, από όποιε αλληλευτικές συμφωνίες και αν δεσμεύεται, ασκεί πραγματικά υπεύθυνη και βιώσιμη αλλία. Γιατί ο ίδιος ο αλληλευτικός κλάδος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην ε, μεταβίβαση αυτού του μηνύματος ότι ασκεί την αλλία με βάση τις συμφωνίες, ότι αλλιεύει υπό το άγρυπνο μάτι των παρατηρητών και πληρεί τις προδιαγραφές και τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας ε, που είναι συμβαλόμενο μέρος σε αυτές τις ελληνικές συμφωνίες. Θα ήθελα να γίνει αυτή η προβολή. Σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια τέτοια ενημέρωση προ τι ε, συμβαλόμενε χώρε για να βοηθήσουμε τον Ευρωπαϊκό Αλληλευτικό Στόλο να αποδείξει αυτή τη δέσμευση. Ακόμη και ω προ του βουλευτέ, να φανεί ότι πραγματικά είναι υπεύθυνη η αλληλεία που ασκούμε. Τελευταία, κυρία Πατράου Σα ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απορρέει από αυτά που ακούσαμε. Τα πρωτόκολλα αυτά περιλαμβάνουν κάποια γενναιόδωρα ποσά χρηματικής αντιπαροχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που η αλληλευτική στόλη και η αλληλευτική προσπάθεια είναι μικρής εμβέλειας. Υπάρχει δυνατότητα διεύρυνση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αύξηση αυτής της αλληλευτική παρουσίας, γιατί είναι εμφανές το ενδιαφέρον της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, να προσθέσει ένα ακόμη γρηγρή σε αυτή την αλληλευτική ζώνη. Υπάρχει λοιπόν έκδηλο και ζωηρό ενδιαφέρον της Πορτογαλίας, για παράδειγμα, που μάλιστα ελίευε στο παρελθόν και έλειπε ένα γρηγρή και έτσι δεν μπορούσε να ελίευσει. Τώρα έχουμε δύο ε, γρηγρή και ενδιαφέρον. Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης ε, του αλληλευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη ζώνη αυτή. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω στην κυρία Πατράου Νέβες ότι κανένα πορτογαλικό γρηγρή δεν είχε δικαίωμα αλλήλευση στη ζώνη αυτή με βάση το προηγούμενο πρωτόκολλο. Και το αίτημα της Πορτογαλίας υπευλήθη δυστυχώς εκπρόθεσμα. Άλλωστε, δεν, το αίτημα της Πορτογαλίας αφορούσε την ευρύτερη ζώνη, όχι την οικονομική αποκλειστική ζώνη της Μικρονησίας. Η καλύτερη λύση είναι στην ανανέωση της συμφωνίας με το Κυριμπάτι. Εκεί θα μπορούσε να υποβάλει επίσημα και εμπρόθεσμα το αίτημα της η Πορτογαλία. Έτσι θα μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα με το πορτογαλικό γρηγορή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλεξάνδρου για να μας δώσει τις ε, εξηγήσεις. Oui, merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω γιατί παρουσιάσατε έτσι πολύ ζωηρά ε, τα, τις λεπτομέρειες αυτού του νέου πρωτοκόλλου που συμπεριλάβαμε πέρσι το μήνα Μάιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ αντικειμενική η παρουσίαση του ιστορικού των λόγων για, τον οποίο, για τους οποίους ε, δεν ε, εφαρμόστηκε το τελευταίο πρωτόκολλο. Πριν ε, να απαντήσω στις ερωτήσεις, τις πολύ σωστές των συναδέλφων σας, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα διαφορετικό σημείο του πρωτοκόλλου, δηλαδή τη σαφή διάκριση μεταξύ των καταβεβλημένων ποσών ε, ε, για τις άδειες και για την ε, υποστήριξη του κλάδου. Πρόκειται για τροποποιήσεις που σιγά σιγά προβλέψαμε όταν ξεκίνησε η συμφωνία το 2010. Ε, πρόκειται για ποσά τα οποία δεν είναι πολύ σημαντικά, αλλά ο αντίκτυπος ε, της διάκρισης που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα επιτρέψει σε κάθε περίπτωση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναστείλει τις ε, πληρωμές ε, του τμήματος της υποστήριξης του κλάδου όταν η υποστήριξη αυτή δεν πληρεί τους ε, στόχους. Πρόκειται λοιπόν για μια ποιοτική αξιολόγηση η οποία είναι άνευ προηγουμένου αν συγκρίνουμε με την κατάσταση που επικρατούσε στις συμφωνίες συνεργασίας στο παρελθόν. Ένα ακόμη ε, θέμα το οποίο έθεσαν ε, πολλοί συναδελφοί σας στις ερωτήσεις τους είναι για ποιο λόγο το προηγούμενο πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε. Κάποιοι μίλησαν για μη σεβασμό των διατάξεων του προηγούμενου πρωτοκόλλου. Θα ήθελα να μιλήσω, θα προτιμούσα να μιλήσω για μη εφαρμογή. Και ο λόγος είναι ο εξής. Υπήρχε ένα μπλοκάρισμα ε, στις, ε, στην επικοινωνία με τις ε, ομόσπονδες πολιτείες της Μικρονησίας, οι οποίοι μας είχαν δώσει έναν λογαριασμό που δεν δεχόταν ευρώ. Οπότε εκεί υπήρξε ένα ε, μπλοκάρισμα της όλης διαδικασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε το πρώτο τμήμα του ποσού ε, του ετησίου ε, για το προηγούμενο πρωτόκολλο και οι πλειοκτήτες πλήρωσαν τις προκαταβολές. Όταν λοιπόν χρειάστηκε να ξαναγίνουν διαπραγματεύσεις ε, με τις ε, ομόσπονδες πολιτείες της Μικρονησίας, ο στόχος μας ήταν να ανακτήσουμε τα ποσά που είχαν καταβληθεί, αλλά που δεν ήταν αντικείμενο αλλιευτικών δυνατοτήτων ε, που είχαν δοθεί από τις ε, Ομόσπονδες Πολιτείες Μικρονησίας και γι' αυτό ακριβώς το άρθρο 1 του πρωτοκόλου γίνεται μια σαφής αναφορά σε μείωση ετήσια 19.000 ευρώ επί του συνολικού θεωρητικού ποσού ε, της ε, καταβολής ε, πληρωμών. Υπάρχει λοιπόν μία αφαίρεση ενός ποσού που θα γίνει κατά τη διάρκεια των τριών ετών του πρωτοκόλου για να καλυφθεί το ποσό των 559.000 ευρώ που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου πρωτοκόλου αλλά ε, που τελικά δεν ε, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο συγκεκριμένο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, χρειάστηκε επίση να δούμε τι θα γίνει με τα χρήματα που είχαν δώσει ω προκαταβολή οι πλειοκτήτε. Ε, στο, στο παράρτημα συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1 τμήμα 2 σημείο 3, σημείο 3α αναφέρεται ότι τα σκάφη που είχαν, είχαν καταβάλει προκαταβολές στο πλαίσιο του προηγούμενου πρωτοκόλου ε, δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τις προκαταβολές για το πρώτο έτος του νέου πρωτοκόλου. Δηλαδή, ο στόχο μας που ήταν να εξασφαλίσουμε αυτά τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί, τα ποσά που είχαν ήδη ε, καταβληθεί, ε, έγινε, ε, υλοποιήθηκε όντω και είναι κάτι το οποίο δέχθηκαν και οι αρχές των ομόσπονδων Πολιτείων της Μικρονησίας. Ήταν άλλωστε μία απαραίτητη προπόθεση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αν αυτό δεν γινόταν αποδεκτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσει. Λοιπόν, αυτός ο στόχο λοιπόν καλύφθηκε. Επιτρέψτε μου τώρα, κυρία Πρόεδρε, να προσπαθήσω να σας απαντήσω με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματα που ετέθησαν από τους συναδέλφους σας. Ε, έγινε αναφορά σε περιορισμένη παρουσία του αλευ... Ευρωπαϊκής Ένωσης, του αλευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, στην ανοιχτή ε, θάλασσα, ε, σε σχέση με τις τρεις συμφωνίες ε, με του, τα, τους, ε, το, τους νήσους Σολομόντος, το Κυριμπάτι και τις ομόσπονδες πολιτείες της Μικρονησίας. Ήταν συμβολική η παρουσία που μας δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε με την παρουσία μας σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο της, ε, και στο πλαίσιο της Επιτροπής Δυτικού Ειρηνικού. Άλλωστε και εσείς συμμετείχατε στις εργασίες ε, της, ε, της ετήσιας συνεδρίασης της WC PFC και γνωρίζετε το κλίμα, το δύσκολο υπό το οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Ε, ξέρετε πολύ καλά ε, ότι ο αληθινός στόλος της Ένωσης γίνεται ε, στόχος ιδιαίτερης, ιδιαίτερων επικρίσεων, παρά το γεγονός ότι οι άλλοι στόλοι είναι πολύ πιο επιθετικοί. Και επίσης μας ε, λένε ότι δεν έχουμε ε, εκπληρώσει τα καθήκοντά μας ε, ως τώρα, κάτι το οποίο είναι πολύ αποθαρρυντικό, γιατί πρέπει επιτέλους να κατακριθούν να κατακριθούν και οι άλλοι εταίροι ε, γιατί αυτό που γίνεται είναι ουσιαστικά κατηγορείται μόνο στο όλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά αυτοί που καταγγέλουν τις ε, δραστηριότητες του αλευτικού στόλου σιωπούν όταν πρόκειται για άλλους στόλους. Οπότε προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας ε, στο πλαίσιο της δικής μας αντιπροσωπεία ε, στην Επιτροπή αυτή για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε καλύτερα τι συμβαίνει διμερώς με τις ε, τρεις αυτές χώρες αλλά και τι γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο WC-CPFC. Λοιπόν, είχε λοιπόν να ζητήσει Είχε λοιπόν ζητηθεί να ενισχυθεί η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στη συγκεκριμένη επιτροπή ε, και σε ορισμένες άλλες επιτροπές του ειρηνικού για να μπορέσει να ανταποκριθεί, να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις ε, που υπήρχαν. Και εσείς κυρία Πρόεδρε θέσατε ένα ερώτημα σε σχέση με την στάση ε, των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας, δηλαδή κατά πόσο το κείμενο του νέου πρωτοκόλλου έχει επικυρωθεί. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, ε, παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο, που είναι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο των Ομόσπονδων Πολιτειών Μικρονησίας. Παρουσιάστηκε λοιπόν το κείμενο και θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και το συντομότερο δυνατόν για να ξέρουμε κατά πόσο ε, εγκρίθηκε το κείμενο που υπευλήθηκε αν τελικά επικυρώθηκε το πρωτόκολλο. Ούτως ή άλλως, όταν ε, κάναμε τις ε, διαπραγματεύσεις με την Μικρονησία τον περασμένο Μάιο, υπήρξε μια σοβαρή βούληση από την ε, εκτελεστική εξουσία της Μικρονησίας για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, να συναυθεί ένα νέο πρωτόκολλο και το νέο αυτό πρωτόκολλο να εφαρμοστεί ορθά. Τώρα, κάτι για τους παρατηρητές. Έχουμε προβλέψει ε, στο πρωτόκολλο αυτό την ε, πληρωμή παρατηρητών 1500 ε, ευρώ και αυτό σύμφωνα με τις συστάσεις της WCPFC. Στα φινελιευτικά όμως και στα γρηγρή. Ε, ήταν όμως ένα από τα προβλήματα των διαπραγματεύσεων. Ε, οι αρχές της Μικρονησίας, ε, που είναι και κυρίαρχες αρχές όταν γίνονται διαπραγματεύσεις με έναν άλλον εταίρο, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για οποιονδήποτε άλλο, επέμειναν να εφαρμοστεί ομοιόμορφα γενικά σε όλα τα σκάφη που αλλιεύουν στην ζώνη της Μικρονησίας να υπάρχει αυτή η εισφορά. Σε σχέση λοιπόν με το πρωτόκολλο το προηγούμενο υπάρχει μία ε, υπάρχει μια επέκταση των πληρωμών αυτών. Είναι, ε, πάση περιπτώσει, είναι επιπλέον κόστος ε, ε, των παραγαδιάρικων, αλλά ο σκοπός είναι να ενισχυθεί και να δείξει σε όλους, σε όσους, στους παράνομους ποια είναι ουσιαστικά η ε, δράση των παραγαδιάρικων αυτών ε, ε, χάρη στην παρουσία παρατηρητών της Μικρονησίας. Κάτι ακόμη σε σχέση με αυτά που ρώτησε η κυρία Πατραών έβεσε για το αίτημα της Πορτογαλίας. Συγγνώμη, αλλά το αίτημα αυτό της Πορτογαλίας έφτασε στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση, μετά τη σύναψη του πρωτοκόλου. Εμείς είμαστε ευέλικτοι αν ε, υπάρξουν ε, σκάφη που δεν ε, εκμεταλλεύονται πλήρως τις αλληλευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο. Υπάρχει ένα αίτημα της Πορτογαλίας το οποίο μπορούμε να, μπορούμε να καλύψουμε. Όμως θα ήθελα να ενθαρρύνω την Πορτογαλία να το αναφέρει αυτό στις επόμενες διαπραγματικές ε, με τα νησιά Κυριμπάτη. Ε, στο πλαίσιο της στρατηγική μας ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε κάποιες αλλιευτικές δυνατότητες επιπρόσθετες για να καλύψουμε το πορτογαλικό αυτό Προσπάθησα να είμαι σύντομος αλλά και περιεκτικός, πλήρης. Αν κάποια ερώτηση ξέχασα, παρακαλώ να μου το επισημάνετε. Ευχαριστώ. No, ε, gracias. Ε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Και συμφωνώ με τα σχόλιά σας. Έχω μία αμφιβολία για τους παρατηρητές. Νομίζω ότι υπάρχει μία μικρή αντίφαση στο πρωτόκολλο για το θέμα αυτό, αλλά θα... ας μην σταθούμε περαιτέρω. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό όμως είναι να μάθουμε αν το Κογκρέσο των Ομόσπονδων Πολιτειών Μικρονησίας θα κυρώσει το πρωτόκολλο. Γιατί αν δεν το κυρώσουν οι βουλευτέ τη Μικρονησία, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα να μα ενημερώσετε για την πορεία αυτή τη διαδικασία. Γιατί, αν δεν κάνω λάθο, τώρα θα πρέπει να ε, συνεδριάζει το Κογκρέσο. Φαντάζομαι θα κρατήσει κανένα μήνα αυτή η ε, συνεδρίαση, γιατί θα έχουν πολλέ εκκρεμότητε, φαντάζομαι. Αυτό είναι το μόνο που μα ενδιαφέρει, να ενημερωνόμαστε για την πορεία τη διαδικασία και το κατά πόσο θα κυρώσει το Κογκρέσο τη Μικρονησία το πρωτόκολλο αυτό. Εγώ ήδη υπέβαλα την έκθεση. Μπορούμε στην επόμενη συνεδρίαση του Μαρτίου να το ξαναδούμε και να ψηφίσουμε στην συνεδρίασή μας του Μαΐου, ώστε να περάσει στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ολοκληρώσαμε το σημείο 5. Ευχαριστούμε κύριε Αλεξάνδρου που ήρθατε στη συνεδρίαση και να μας ενημερώσετε. Περνάμε στο σημείο 6 που αφορά το πρόγραμμα στήριξης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Πατράο Νέβες και θα μας εξηγήσει πώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την Επιτροπή Μεταφορών ως προς την ε, αμφισβήτηση επί της ουσίας που υπάρχει. Θα ήθελα καταρχήν να σας παρουσιάσω κάποια διαδικαστικά ζητήματα για την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή ανατέθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών, όπως ξέρετε, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας. Και η δική μας αλληλευτική ε, επιτροπή ανέλαβε την εκπόνηση της γνωμοδότησης. Η Επιτροπή Αλίας όμως θεώρησε ότι για το θέμα αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί ως συνδεδεμένη επιτροπή με την Επιτροπή Μεταφορών και εκθέσαμε και τα επιχειρήματά μας για το αίτημα αυτό. Όλοι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ο σχετικός κανονισμός στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι θα πρέπει να ευθύσουμε μια οριζόντια, ολιστική, σφαιρική προσέγγιση για τη θάλασσα. Αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται μια τέτοια ολιστική προσέγγιση, σφαιρική, και αντίστοιχη σφαιρική προσέγγιση θα πρέπει να υιοθετήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θάλασσα. Άρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιτρέψει δύο επιτροπές ε, να προσεγγίσουν αυτό το θέμα ως αρμόδιες κατ' ουσία και να μην αφήσουμε μόνο την Επιτροπή Μεταφορών να επιληφθεί αυτού του θέματος. Γιατί χρειαζόμαστε μία κατακόρυφη ε, σφαιρική και συγκροτημένη προσέγγιση για το θέμα της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής. Άλλωστε υπάρχει ήδη το προηγούμενο της ενισχυμένης συνεργασίας και νομίζω ότι και στην περίπτωση αυτή συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε, συνεργασίας των δύο επιτροπών για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Άλλωστε ο κανονισμός περιλάμβανε και διάφορα σημεία που έκαναν προφανή την ε, επί της ουσίας αρμοδιότητα και της δικής μας Επιτροπή. Για παράδειγμα, το άρθρο 2, εδάφιο Δ, το άρθρο 3, ολόκληρο το άρθρο 3, σημείο 1 ιδιαίτερα, αλλά και το σύνολο του άρθρου 3, παράγραφος 2, εδάφιο Β, συνηγορούν προς την αρμοδιότητα της Επιτροπής. Εκεί μιλούμε για την ε, βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και μιλούμε για συστημική προσέγγιση που είναι πολύ σημαντική για τον αλληλευτικό κλάδο. Τα δύο αυτά άρθρα, 2 Δ και 3 δβ αναφέρονται στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η Επιτροπή Αλίας ως προς την σύναψη ελευθερικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Οπότε, υπάρχει επιχειρηματολογία που θεμελιώνει τη διεκδίκησή μας να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Μεταφορών για την διεκδίκηση της καθήλια αρμοδιότητας με βάση το άρθρο 50 του κανονισμού. Κινητοποίησαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε την απόφαση. Υπήρξε μια ανταλλαγή αλλογραφίας και μάλιστα πριν από λίγο έμαθα ότι αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για τη 15η Φεβρουαρίου, κάτι που ήταν απροσδόκητο μάλλον, γιατί εμείς περιμέναμε μετά την ε, τελευταία μας επιχειρηματολογία και παρουσίαση του θέματος η διάσκεψη των Προέδρων θα είχε δεχτεί την πρότασή μας και τελικά διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής η Επιτροπή Μεταφορών μένει αμετακίνητη και αδιάλακτη. Δεν διευκολύνει καθόλου το αίτημά μας ε, να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα η διάσκεψη των Προέδρων πρότεινε αναβολή της απόφασης ως προς τη σύσταση που κάναμε εμείς. Οπότε η διαδικασία μέχρι στιγμής δεν μας δημιουργεί και μεγάλη αισιοδοξία, αλλά είμαι βεβαία ότι και η Πρόεδρος θα έχει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή. Προς το παρόν έτσι έχει η κατάσταση, εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες, εν αναμονή βέβαια της απόφασης, και εμένοντας στο έτοιμά μα ε, να θεωρηθούμε ω συνδεδεμένη επιτροπή, μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών. Ο κανονισμός προβλέπει ένα σύστημα υποστήριξη για την εμβάθυνση της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής που εξασφαλίζει την απαραίτητη νομική βάση για τη χρηματοδότηση ε, συναφών δραστηριοτήτων τη εφαρμογή τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Προβλέπεται χρηματοδότηση για να καλυφθούν ε, τα έξοδα από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 και μάλιστα η χρηματοδότηση έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010, οπότε έχει, νόημα να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία και να τη συνεχίσουμε. Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της έκθεσης αυτής και του κανονισμού αφορά κάποια πειραματικά σχέδια, σεμινάρια, συνέδρια, μελέτες, προγράμματα συνεργασίας, ενημέρωση του κοινού, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, επιτήρηση και δρομολόγηση πληροφοριών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον κανονισμό είναι απολύτως απαραίτητες για να συγκεκριμενοποιήσουμε τις, ε, τους προσανατολισμούς της έκθεσης πρόοδου που Μα υπευλήθη τον Οκτώβριο του 2009. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική παρουσιάστηκε ως ε, σημαντική πολιτική που θα επιτρέψει την ανάπτυξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προ... προκάλεσε τεράστιες προσδοκίες, πολύ ψηλές προσδοκίες. Δυστυχώς ε, προς το παρόν έμεινε σε φάση ακινησίας για να η επιβράδυση, για να μην πω αποτελμάτωση, αποτελμάτωσης και θα πρέπει επουδενή να επιτρέψουμε αυτή η πενιχρή με χρηματοδότηση αλλά σημαντική να καθυστερήσει περαιτέρω, γιατί μια περαιτέρω καθυστέρηση αυτής της έστω και μικρής χρηματοδότησης ε, θα κινητοποιήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες που εξακολουθούν να κρατούν μέχρι στιγμής ενεργό την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Και από το 2013 θα επιτρέψουν μια πραγματική πλήρη εφαρμογή αυτής της θαλάσσιας πολιτικής. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό ποσό αυτής της πολιτικής που είναι πραγματικά πενιχρός υπολογισμός, το απολύτως απαραίτητο για να διατηρηθούν αυτές οι δραστηριότητες από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 και θα ε, χορηγηθούν από τη στήλη 2 του κοινοτικού προϋπολογισμού αυτά τα ποσά. Πρόκειται για μια στήλη που αναφέρεται ως περιθώριο αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπάρχοντα κονδύλια που μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, καταμεριστεί. Αυτά τα 50 εκατομμύρια βέβαια Αυτά 50 εκατομμύρια δεν θα βγουν από κανένα αλληλευτικό ταμείο. Είναι πενιχρός αυτός ο υπολογισμό των 50 εκατομμυρίων, αλλά χρειάζεται. Θα ήθελα να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένες προτάσεις τώρα του κανονισμού. και πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Το άρθρο 8 του κανονισμού μιλά για τον προσδιορισμό της προέλευσης του, της χρηματοδότησης, γιατί αναφέρεται η χρηματοδότηση, αλλά δεν ξέρουμε από πού θα προέλθει. Και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έλαβα εγώ, αν επιβεβαιωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να προσδιορίσουμε την πηγή της χρηματοδότησης, την προέλευση της χρηματοδότησης. Μια άλλη πρόταση τροπολογίας τροποποιεί το άρθρο 13 που μιλά για τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι απλώς συμβουλευτική, όπως λέει και το όνομά της. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επιρροής ή παρέμβαση στις εξουσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι αρμοδιότητε της για τη διαμόρφωση των αιτήσεων προσανατολισμών και κατευθυντήριο γραμμών για την εκτέλεση, την υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Νομίζω ότι έχει νόημα να ενισχύσουμε και τη θέση και τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής. Αναφέρεται ως ρυθμιστική μια αριθμιστική επιτροπή που θα είναι μια επιτροπή με ενισχυμένε αρμοδιότητες. Η ισχύουσα μέχρι στιγμή αριθμιστική επιτροπή θα καταργηθεί και μιλούμε πια για ένα νέο μοντέλο δράσης που προϋποθέτει και μια διαδικασία εξέτασης αντίστοιχη με αυτή που ισχύει σήμερα για την Ρυθμιστική Επιτροπή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν το καταστατικό και τις αρμοδιότητες της συμβουλευτική Επιτροπής και να επιτρέψουμε μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβαση σε θέματα ολοκληρωμένη θαλάσσης πολιτικής. Και να θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημείο αυτό. Θα ήθελα να μα εξηγήσει καλύτερα ποια είναι η εναλλακτική λύση ως προς τη Συμβουλευτική αυτή Επιτροπή. Αυτή η examination procedure, αυτή η διαδικασία εξέταση που αναφέρεται, σε τι ακριβώ αντιστοιχεί. Σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε τώρα. Ελήψη απόφασης ε, ως προς το αίτημά μας για να γίνουμε συνδεδεμένη επιτροπή έχουμε ως χρονοδιάγραμμα για την ε, υποβολή της έκθεσης 15η Μαρτίου. Αλλά ακόμη δεν έχουμε λάβει, απόφαση, δεν έχουμε λάβει απάντηση ως προς το αίτημά μας. Οπότε δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατράου. και κυρία Ρέιμερς. Yeah. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω σαφώς τους συναδέλφους μας. Πρέπει να θεωρούμε την αλληλεία ως ισότιμο μέλος στην ολοκληρωμένη πολιτική, διότι έτσι είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσουμε την επάρκεια τροφίμων, η οποία αναφέρεται βεβαίως στον κανονισμό, τον αντίστοιχο κανονισμό, όπως και στον αγροτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ισότιμος εταίρος και επίσης ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Θέλω να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική για την περιφέρειά μου, διότι εμείς ε, ναι, λειτουργούμε ως κράτος μεταξύ δύο θαλασσών, Ατλαντικού Βορείου και έτσι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα διαφορετικά αιτήματα και τις διαφορετικές πραγματικότητες. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουμε κι εμείς. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Also... Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία για αυτή την γνωμοδότηση, διότι αν θεωρήσετε ότι η Επιτροπή Μεταφορών είναι η η αρμόδια, τότε είναι επί της ουσίας ε, και τα θέματα τα οποία καλύπτονται από την, ε, την τον κανονισμό αυτόν, ε, είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς, εάν λάβετε υπόψη τις μεταφορικές δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και την, ε, τα προβλήματα με τα καύσιμα, το πετρέλαιο, πρέπει και η Επιτροπή Ενέργειας να έχει έναν λόγο ε, στο νησί Ταϊρή, στη δυτική ακτή της υπάρχει ένα αιωλικό πάρκο και το επισκέφθηκα και μου είπαν ότι έχουν πρόγραμμα να επεκταθεί αυτό το αιωλικό πάρκο ε, και να ε, καλύψει μια περιοχή όπως όλη η Σκοτία. Θα έχουμε λοιπόν στο μέλλον πιστεύω τεράστιες ε, offshore, τεράστια offshore αιωλικά πάρκα και γι' αυτό θα πρέπει και ε, να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα της αλίας που θα παρουσιαστούν σε αυτές τις περιφέρειες όταν εγκατασταθούν αυτές οι τεράστιες αναμογεννήτρες. Ε, υπάρχουν τρομερές πιέσεις από απόψεως περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Πολλές φορές τα προγράμματα αυτά δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την τοπική αλία και λένε θα πάει κατά διαβόλου, τι μας νοιάζει εμάς. Λοιπόν, ε, όλες αυτές, ε, όλοι αυτοί οι τομείς, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, ε, έχουν τεράστιες επιπτώσεις πάνω στην αλληλεία και την αλλιευτική κοινότητα. Γι' αυτό είναι πρωταρχική σημασία να υπάρχει το καθεστώς της ενισχυμένης συνεργασίας με μας. Ευχαριστώ κύριε Γκρομπάρτσικ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, προσθέτοντας σε όλα αυτά που ακούσαμε, να πω ότι η ιστορία τελικά επαναλαμβάνεται. Και πέρυσι είχαμε έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ακόμη και η επιλογή της διαδικασίας αυτής της έκθεσης δεν μας γέμιζε με αισιοδοξία, γιατί η Επιτροπή Μεταφορών κρίθηκε αυτή η έκθεση ως ε, ε, δευτερεύουσα. Και επειδή χαρακτηρίστηκε ως μη ουσιαστική αυτή η έκθεση, χρειάστηκε να συγκεντρώσουμε 70 υπογραφές για να καταθέσουμε τροπολογίες, ακριβώς επειδή χαρακτηρίστηκε σήμαντη ουσιαστικά αυτή η Επιτροπή. Τελικά, από όλε τι τροπολογίε που καταθέσαμε, μόνο μία λήθη υπόψη. Αυτό δείχνει ποια είναι η προσέγγιση τη Επιτροπή Μεταφορών ω προ τα θέματα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και διαχείρισης της θάλασσας και εκμετάλλευσης. Μιλούμε πολύ συχνά ότι χάνουμε τα σκάφη μας που προτιμούν κινέζικη σημαία ή άλλες σημαίες ευκαιρίας. Μιλούμε επίσης για φορολογικούς ε, παραδείσους, για θέματα ανάγκης ε, ανασύστασης ε, και αναζωογόνησης ε, του τομέα των αυπηγείων. Φαίνεται ότι όλος αυτός ο κλάδος ε, της θαλάσσιας οικονομίας εξωθείται στην περιθωριοποίηση. Εγώ προσπάθησα στην ομάδα μου να κάνω μια ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία αυτού του τομέα και πόσο σημαντικό είναι να κριθεί αρμόδια η Ελευτική Επιτροπή για να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη γνώμη του σε θέματα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και οικονομίας. Γιατί η θαλάσσια οικονομία είναι μια, ένας κλάδος που δυστυχώς δεν είναι αρκετά αναπτυγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντρεβαρέα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Πατράου. Φαίνεται ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν είναι το τομεακή, αλλά οριζόντια και επηρεάζει και διαφέρει πολλές πολιτικές της Ένωσης, γιατί υπάρχει διασύνδεση των πολιτικών, γιατί η αλλήλεια είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της θαλάσσιας πολιτικής και θα πρέπει να προβλέψουμε και ένα προϋπολογισμό που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες, που θα μας επιτρέπει να συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και να προβαίνουμε σε και σε πολιτικές αναλύσεις. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί μπορεί να επηρεάσει και να έχει παρενέργειες και σε άλλες καταστάσεις, αλλά και να επηρεάσει αρνητικά αλληλευτικούς πληθυσμούς. Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εξασφαλίσουμε συναρμοδιότητα με άλλες επιτροπές και διαδικασίες συναπόφασης και η Επιτροπή Ενέργειας είναι σημαντική, όπως είπε ο κύριος Στίβενσον, γιατί υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ε, οικονομικών κινήσεων στη θάλασσα. Έχουμε νέες μορφές βιομηχανικής παραγωγής, για παράδειγμα, που θα χρειαστούν μελέτες επιπτώσεων και θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό λοιπόν πιστεύω θα πρέπει να είναι το σημείο αφετηρίας μας και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο ειδικό βάρος της Επιτροπής μας για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό της θαλάσσια ολοκληρωμένη πολιτικής. Άλλωστε, ο τομέας αρμοδιότητάς μας κινείται σε αυτό το περιβάλλον που είναι το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο κύριο Μίλαν. Και Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάνω από ένα, ε, περισσότερα προβλήματα. Υπάρχει ένα θέμα αρχής. Ενώ συμφωνώ με την εισηγήτρια θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά τη μόνο τη διαδικασία συνεργασίας. Έχει και πολιτική ουσία και αφορά και τον πρόεδρο του σώματος και την επιτροπή μας. Εάν δηλαδή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, σε ποιο πλαίσιο ανήκει. Πού ακριβώς τοποθετείται. Θυμάμαι ότι και παλαιότερα είχαμε ένα πλαίσιο ενισχυμένη συνεργασία, το οποίο κατέληξε στην εφαρμογή του κανόνα 50. Και θα πρέπει να υπεραμεινθούμε τις θέσεις μας έντονα πρέπει να απαιτήσουμε να μας ε, δοθεί ε, μία ε, καθοδήγηση, να λάβουμε, μία, να λάβουμε σαφείς οδηγίες. Διότι εάν 80% των πόρων δεν χρησιμοποιούνται για μεταφορικούς σκοπούς, ακόμα και στην πρόταση της Κομισιόν, και αν το 70% θα καλύψει δύο ουσιαστικούς στόχους, δηλαδή την ε, θαλάσσια βιοπικιλότητα και συναφή μέτρα και την, ε, τον έλεγχο και εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση εποπτεία. Εάν λοιπόν το 70% καλύψει αυτές τις δύο πτυχές, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό αναφέρεται σε έναν μόνο κλάδο, σε έναν μόνο τομέα. Διότι η αλληλεία πρέπει να έχει το δικό της κλάδο επισόρησης και εποπτείας. Ας θυμηθούμε παλιότερα που είχαμε πει να δημιουργήσουμε μία τράπεζα δεδομένων, διότι τότε είχαμε κατά νου ακριβώς αυτό το στόχο καταγραφής όλων των στοιχείων επιθεώρησης ε, έπρεπε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων για όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι λοιπόν μόνο ζήτημα ισχύω ε, το ότι πρέπει να έχουμε έναν πολύ ισχυρό κλάδο και να είμαστε πολύ δυνατοί έναντι ε, της Επιτροπής Μεταφορών και γι' αυτό το λόγο να ζητάμε ε, ενισχυμένη συνεργασία. Πιστεύω ότι υπάρχει και η πολιτική πτυχή που δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Διαφορετικά ε, δεν θα είχα αυτή τη γνώμη. Θέλουμε μία ισχυρή πολιτική, να είμαστε δυνατοί, έτσι ώστε να είμαστε και επιτυχείς όταν παρουσιαστούμε στην Ολομέλεια με τις τροπολογίες μας. Και εν πάση περιπτώσει να μην αγνοηθούμε, να μην είμαστε εκτός αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν λοιπόν στον ε, κανονισμό ως έχει πάρα πολύ σαφή όρια. Καταρχάς, πρέπει να εφαρμοστούν, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στου πίνακες του κανονισμού. Υπάρχει υπερβολική ελευθερία ερμηνείας, διότι μα είπε η Κομισιόν ότι αυτά τα παραρτήματα και οι πίνακε δεν αποτελούν μέρος της γνωμοδότησης, ε, επειδή αφορούν βασικά διαδικασίε μεταφορών. Οπότε, η διαχείριση του τομέα μπορεί να υπονομεύσει τη, τα πολιτικά επιχειρήματα, τους πολιτικούς στόχους. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε ένα ουσιαστικό κείμενο και να μην αφήσουμε τους πίνακες, τα παραρτήματα. Πιστεύω ότι αποτελούν μέρος της ουσίας, διότι όπως σας είπα περιλαμβάνει πολιτικά στοιχεία. Η εφαρμογή του εγγράφου, του κειμένου αυτού έχει πολιτικές πτυχές. Δεύτερον, πιστεύω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ στενή ερμηνεία όσον αφορά την, τον προορισμό των πόρων. Πού δηλαδή θα καταλήξει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Περιορισμένη οπτική, περιορισμένη οπτική ερμηνεία. Ε, Πού θα καταλήξει τελικά. Ε, ας μην ε, περιοριστούμε μόνο στην, στις ακτές, δηλαδή ότι μόλις η θάλασσα κουμπίσει γη, σταματάει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ότι αφορά και καλύπτει μόνο τις παράκτιες περιοχές έχει και άλλες επιπτώσεις. Είναι ευρύτερη πιστεύω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, επεκτείνεται και πέραν από τις καθαρά ε, και μόνο παράκτιες περιοχές. Εάν εξετάσετε, αν δείτε τις απορρίψεις και το περιεχόμενο σε διοξίδιο του θείου, ε, τι επιπτώσεις έχουν οι απορρίψεις λοιπόν αυτές, όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στους, στα ποτάμια και στα εσωτερικά υδατά, θα δείτε ότι οι επιπτώσεις ε, είναι ευρύτερε. Σκεφτείτε την ε, θαλάσσια ισορροπία στην Αδριατική και πώς τι επιπτώσεις έχει στην Ιταλία η αυξημένη θαλάσσια μόλι, ρήπανση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε να λειτουργεί η πολιτική αυτή βάσει ενός σωστού προγράμματος ελέγχου και παρακολούθησης ένας μεγάλος και να λάβουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και των ε, ποτάμιων νεκρών. Παραδείγματο χάρη ο ποταμός ε, Πο στην Ιταλία μέσω του οποίου χύνονται τεράστιες ποσότητες, ε, ο <laughs> συγγνώμη, μέσω του οποίου χύνονται τεράστιες ποσότητες βλαβερών ουσιών στην θάλασσα. Πιστεύω λοιπόν ότι αντί να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση με την Επιτροπή Μεταφορών, δεδομένου ότι μια διαπραγμάτευση μπορεί να οδηγήσει σε ήττα ή σε νίκη, θα πρέπει να δούμε εμείς την ενισχυμένη θέση μας καταρχάς. Και δεύτερον, αν δεν θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας οι ενδιαφερόμενοι, να αρνηθούμε να συντάξουμε γνωμοδότηση. Γενικά, θα πρέπει οι βασικές αρχές να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Και τέλος, στην, στον αρχικό τίτλο γίνεται μία παραμπομπή στο 74 και 77 της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτά τα δύο άρθρα της Λισαβόνας αναφέρονται στον τομέα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. από ό,τι καταλαβαίνω αφορά ακριβώς τα δικαιώματα πρόσβασης ε, στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν η παραπομπή σε αυτά τα δύο άρθρα να διαγραφεί. Τελείως. Και να μην, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να κατευθυνθούν οι πόροι μας σε κεφάλαια και τίτλους που δεν τους επιθυμεί διόλου το Κοινοβούλιο. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω ε, την συγκεκριμένη και πιστεύω ah, ότι πρέπει όλοι να έχουμε μια ισχυρή θέση, διότι η πολιτική μεταφορών αποτελεί ένα μέρος της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας ε, πολιτικής. Ε, στο παρελθόν, λέει η κυρία Ρόνταστ, είχαμε πει ότι δεν πρέπει να μείνουμε ε, εκτός συζητήσεων όταν συζητούνται παρόμοια θέματα σε διαφορετικές επιτροπές. Πρέπει να συμμετέχουμε εμείς ιδίως σε θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή ε, είναι, είναι, συζητιούνται διεθνώς. Είναι θέματα που αφορούν ε, όλους. μιλάμε για μια ολοκληρωμένη πολιτική, καλύπτει πάρα πολλά θέματα, επίσης και χωροταξικά. Θα πρέπει κάποια στιγμή να εποφεληθούν από τις, ε, τους ωκεανούς ε, και τα, τα, θαλάσσια περιβάλλον. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε μια θαλάσσια πολιτική μόνο στην αυσιπλοεία, ε, στις μεταφορές. Αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Είμαι λοιπόν βέβαιη ότι πρέπει οπωσδήποτε, έχουμε το δικαίωμα δηλαδή να συμμετάσχουμε ισότιμα σε όλο αυτό το διάλογο. Μάλιστα θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε η, Επιτροπή επί της ουσίας. Ε, ε, το μόνο που, θα δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να αποσυρθούμε και να χάσουμε έδαφος. Danke, Κύριο Σκούν, ευχαριστώ. Η συγγήτρια ακριβώ ξεκίνησε από τη σωστή θέση. Μπορούμε να συζητάμε πιο και να πούμε ότι τα λιευτικά σκάφη ε, συμμετέχουν εξίσου στις ε, διεθνεί θαλάσσιε μεταφορές και στις ε, μεταφορέ στα εσωτερικά ύδατα. Πρέπει τα αλλιευτικά ε, σκάφη να ε, ακολουθούν ακριβώς τους ίδιους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που είναι σωστό, πρέπει να ενεργούν και να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως και η Διεθνής Ναυτιλία. Ωραία και καλά όλα αυτά. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, πρέπει να λάβει υπόψη και την οικολογική θαλάσσια διακίνηση. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ακριβώς οι μεταφορές εκείνες οι οποίες έχουν τις λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου ανατόνο και αναεπιβάτη. Εάν εξετάσουμε τις κινήσεις των αλλιευτικών μας ε, στόλων θα έλεγα ότι οι οικολογικές επιβαρύνσεις είναι σταθερές ή, και, ή βαίνουν προς τα κάτω, είναι ευθύνωσες. Οι αυξημένες λοιπόν θαλάσσιες μεταφορές στη, Βόρεια Θάλασσα, στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο έχει σαφώς επίπτωση στους πόρους, στους διαθέσιμους πόρους μας. Και ο συνάδελφος από τη Σκωτία το είπε ξεκάθαρα εμείς δεδομένου ότι όλο και περισσότερο γίνεται εκμετάλλευση των θαλασσών είτε με αξιοκαλλιέργειες, είτε με ολικά πάρκα, είτε με άλλους τρόπους, παραδείγματο χάρη ε, αγωγή αερίου ή πετρελαίου περνάνε από, ε, διαμέσου των θαλασσών. Λοιπόν, όλη αυτή η αυξημένη χρήση των θαλασσίων πόρων έχουν σοβαρές επιπτώσεις διεθνώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το δικό μας τομέα πρέπει σαφώς να έχουμε το ίδιο τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή Μεταφορών. Δικαιώματα διαβούλευσης και για λόγους ασφαλείας και για περιβαλλοντικούς λόγους μιλήσαμε για περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου, Επίσης, για λόγους ε, αποβολής του, του, έρματος των ε, σκαφών που επηρεάζει τη βιοπικιλότητα. Άρα, λοιπόν, συμφωνώ με αυτή την ε, προσέγγιση 100%. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου καινούριο και μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η θαλάσσια ολοκληρωμένη πολιτική δεν έχει δική της νομική βάση, ούτε στη συνθήκη, ούτε στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο παράρτημα 7, που είναι το αντίστοιχο με τις, για τις αρμοδιότητες των διαφόρων επιτροπών. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, ο κύριος Καπόλος, που ήταν ο, ο μόνος μαζί με τον κύριο Στίβενσον που ήταν στο Κοινοβούλιο για το, αρμόδιο για το θέμα αυτό, είχαμε υποβάλει μία τροποποίηση του κανονισμού, του παρατήματος 7, για τις αρμοδιότητες των επιτροπών. Και μάλιστα είχαμε διεκδικήσει για την Επιτροπή Αλίας την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Όχι αποκλειστικά, κατά αποκλειστική αρμοδιότητα, αλλά θεωρούσαμε ότι και για μας αυτό το θέμα ήταν πολύ σημαντικό. Βέβαια το θέμα είναι ιδιαίτερα πολιτικό και η Επιτροπή Μεταφορών δεν θέλει να αφήσει και άλλες επιτροπές ε, να συμμετέχουν στο σημείο αυτό ως συναρμόδιες. Εντάξει, συνεργασία ναι, αλλά γιατί κανένας δεν αφισβητεί ότι είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα και για την αλληλευτική πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι αν κάποια επιτροπή ή αν κάποια κοινοτική πολιτική έχει ιδιαίτερη σχέση με την θαλάσσια, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αν υπάρχει μία τέτοια κοινοτική αρμοδιότητα και πολιτική, αυτή είναι η αλία. Οπότε είναι λογικό να έχουμε και την ε, οικοσυστημική ε, προσέγγιση που μας συνδέει άμεσα με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ο ελευτικός κλάδος και η ελευτική πολιτική είναι κατεξοχήν κοινοτική πολιτική. Οπότε αν κάποιος συναρμόδιζε το συντονισμό σε αυτά τα θέματα είμαστε εμείς, η Επιτροπή Αλίας. Πάντως όντως είναι περίπλοκο το ζήτημα και από πολιτική άποψη και σίγουρα δεν θα εγκαταλείψουν ε, τη θέση τους ε, τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Πάντως νομίζω ότι σε θέματα ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής η συμμετοχή μας είναι αναφυσβήτητα. Το θέμα είναι σε ποιο επίπεδο θα φτάσουμε. Το λιγότερο κατά τη γνώμη μου, το ελάχιστο θα ήταν το άρθρο 50. Το σωστό θα ήταν το άρθρο 51 ώστε δύο επιτροπές που είναι άμεσα αναμειγμένες να συνεδριάζουν από κοινού και να συναποφασίζουν. Βέβαια από πρακτική άποψη είναι δύσκολο να εφαρμοστεί το άρθρο 51 και γι' αυτό ακριβώς το άρθρο 51 δεν εφαρμόζεται πιθά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της περιπλοκότητάς του. Είμαι από τους ελάχιστους ε, που υποστηρίζω αυτό το θέμα, γιατί με το που κάνω εγώ ένα βήμα μπρος, με τραβάνε πίσω τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Όχι επειδή έχουν πιο ε, έξυπνη επιχειρηματολογία, αλλά επειδή είναι πολύ ισχυρή η Επιτροπή Μεταφορών. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ενθαρρύνω και να σας παροτρύνω όλους. Είτε κάποια διαβήματα στους ε, συντονιστές ε, των, της Επιτροπής Μεταφορών, είτε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, που είναι σοσιαλιστής. Κάντε ό,τι μπορείτε για να υποστηρίξετε το θέμα μας. Είναι απαράδεκτο η Επιτροπή Μεταφορών για όλα αυτά τα θέματα της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής να έχουμε εφαρμόσει το άρθρο 50, την ενισχυμένη συνεργασία και τώρα που φτάνει ένα στοιχείο που είναι συναπόφαση να αποφασίζει η Επιτροπή Μεταφορών ότι εμείς περιτεύουμε και να διεκδικούν την απόλυτη, αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι τελείως ανεδαφικό το επιχείρημά τους. Βέβαια είπαμε, έχει ισχύ η Επιτροπή Μεταφορών, γι' αυτό και προτάσει τα επιχειρηματά της. Ο κύριος Σίμψον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, συμπαθέστατος άνθρωπος, το μόνο που είπε απαντώντας στην ε, παρατήρησή μου ήταν «Ε, η αλία είναι αλία και οι μεταφορές είναι μεταφορές». Άρα, φως φανάρι, αποκλείεστε εσείς η Επιτροπή Αλίας. Εγώ πάντως θα συνεχίσω τον αγώνα, δεν πρόκειται να καταλήψω. Δεν πρόκειται να παρατηθώ, αλλά το θέμα είναι περίπλοκο. Ό,τι μπορείτε να κάνετε προς τους συντονιστέ, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών είναι ευπρόσδεκτο. Πάντως σίγουρα δεν θα πρέπει να παρατηθούμε, να εγκαταλείψουμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι προς την κυρία Πατράου, μια διαφωνία. Κυρία Μπιλμπάου, μην βιάζετε, θα σας δώσω το λόγο, τώρα μιλάω εγώ. Κύριε Πατράου, στην σελίδα 21, στο σημείο 412 στα ισπανικά, μιλά για την ασυμβατότητα του οικονομικού προγραμματισμού, του δημοσιονομικού προγραμματισμού. Είπατε ότι αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ θα χορηγηθούν από το περιθώριο της δεύτερης κατηγορίας. Στο 412, εκεί που μιλάτε για συμβατότητα του δημοσιονομικού ε, προϋπολογισμού, μιλάτε για ανάγκη αναπρογραμματισμού των, των στυλών του προϋπολογισμού. Άλλο αναπρογραμματισμός, άλλο περιθώριο της κατηγορίας 2. Δεν είναι σωστό λοιπόν αυτό που λέτε ότι τα 50 εκατομμύρια θα βγουν από τα αλλιευτικά κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Οπότε δεν ευσταθεί αυτό που είπατε ότι θα βγουν από το περιθώριο της κατηγορίας 2. Βγαίνουν από το κεφάλαιο αλία, αλίας και τα, τα, από τα ναυτιλιακά. Αν το θέλουν και αυτό οι αν θέλουν αυτό το θέμα η Επιτροπή Μεταφορών, τότε να το χρηματοδοτήσουν από τα κονδύλια των μεταφορών. Γιατί να το χρηματοδοτεί το κεφάλαιο Ελίας. Αν θέλουμε ένα προγραμματισμό, καλύτερα να αναπρογραμματίσουμε τα κεφάλαια Ελίας για αλλιευτικά ζητήματα, για τα θέματα που έχουμε λόγο και όχι για τη θαλάσσια, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που τη διεκδικεί αποκλειστικά η Επιτροπή Μεταφορών, αν τη διεκδικεί να τη χρηματοδοτήσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σα πω μια σχετικά χιδέα παροιμία στα ισπανικά που πραγματικά θα ήταν ε, τα μάμ για την περίπτωση αυτή κουτί, αλλά επειδή είναι κάπως ε, τολμηρή δεν θα σας την αναφέρω. Κυρία Μπιλμπάου, συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπαμε. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά συμφωνώ ότι και η Επιτροπή Αλίας ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα και θα πρέπει να διεκδικήσει την αρμοδιότητά της. Και αυτό θα ήθελα να πω, ότι θα κάνω ό,τι μπορώ μέσω της Επιτροπής ε, Μεταφορών για να προωθήσω το επιχείρημά μας και το έτοιμά μας. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρέμβει εδώ στην εσωτερική συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων επιτροπών. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για να καταφέρουμε ε, οι συνομοθέτες να φτάσουν στη συμφωνία μεταξύ τους το συντομότερο δυνατόν ώστε το συντομότερο δυνατό το 2011 να έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το μέσο που είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση κάποιων δραστηριοτήτων που κατοχυρώνουν και εμπεδώνουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αυτός ο εγκάρσιος χαρακτήρας της ε, ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που επισημάνθηκε είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής. Οπότε οτιδήποτε υπογραμμίζει αυτόν τον, υπογρα... τον εγκάρσιο χαρακτήρα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι ευπρόσδεκτο. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Και η κυρία Πατραονέβες, αλλά και εσείς και άλλοι ομιλητές, αναφέρθηκαν στο θέμα της πηγής της προέλευσης της χρηματοδότησης. Θα ήθελα καταρχήν να σας επιβεβαιώσω ότι αυτό ο προπολογισμό των 50 εκατομμυρίων ευρώ προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο της στήλη 2 των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013. Αυτά τα χρήματα δηλαδή ανήκουν στο ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται για επιπλέον κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αλλά προέρχεται από το δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη πολιτική που ε, χρηματοδοτείται από τη γενική κατηγορία της στήλη 2. Και όταν μιλούμε για ένα προγραμματισμό δεν εννοούμε για ένα προγραμματισμό των αλλιευτικών κονδυλίων, αλλά του συνόλου της στήλη 2. Δηλαδή, κάποια κονδύλια που υπάρχουν στη στήλη 2, στο περιθώριό της όμως, δηλαδή δεν έχουν κατανεμηθεί και άρα δεν ανήκουν σε καμία αλλιευτική ή καμία άλλη πολιτική της Στήλη 2, να δοθούν σε αυτήν την χρηματοδότηση, αντί να μείνουν σε, αυτό το, σε αυτή την δημοσιονομική απαθή ζώνη που είναι το περιθώριο. Επαναλαμβάνω, τα 57 εκατομμύρια δεν θα φερεθούν από τον προϋπολογισμό της αλίας σε καμία περίπτωση. Αλλά ένα μικρό τμήμα των κονδυλίων που βρίσκονται στο περιθώριο της στήλη 2 θα αφιερωθούν στη χρηματοδότηση των μέτρων της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Για τις ερωτήσεις κυρίας Το θέμα των επιτροπών. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την Συμβουλευτική Επιτροπή και όχι Εξεταστική Επιτροπή. Για πολλούς και διάφορους λόγους που θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ο γενικός κανόνας στην επιτροπολογία με βάση τις νέε διατάξεις. Επίση θεωρούμε ότι η πιθανή χρήση της εναλλακτική λύσης, που είναι η Εξεταστική Επιτροπή, αυτή η Εξεταστική Επιτροπή προβλέπεται για συγκεκριμένε περιπτώσει και υπό συγκεκριμένε προποθέσει που δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιε είναι αυτέ οι προποθέσει, Για παράδειγμα, η πρόταση θα πρέπει να έχει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες. Εδώ και λόγω του ποσού, τα 50 εκατομμύρια. Αλλά κυρίως επειδή αυτό το ποσό προέρχεται από ένα ε, δημοσιονομικό περιθώριο εντός των δημοσιονομικών προοπτικών της Ένωσης. Δεν πρόκειται για πρόσθετα δηλαδή κοινοτικά κονδύλια του προπολογισμού. Γι' αυτό και δεν είναι σημαντικές οι δημοσιονομικές συνέπειες και άρα δεν πληρείται αυτή η προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή τη Εξεταστικής επιτροπή είναι η πολιτική ευαισθησία του θέματος. Μέχρι στιγμής, στις συζητήσεις που έγιναν και με τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής, σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε η πολιτική ευαισθησία του ζητήματος. Υπάρχει μάλλον αμέριστη υποστήριξη για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και την εφαρμογή αυτού του πενιχρού προϋπολογισμού για τη δράση της. Οπότε δεν υπάρχει ούτε πολιτική ευαισθησία. Τρίτη προϋπόθεση είναι να πρόκειται για μέτρα ευρεία εφαρμογή. Ούτε και αυτό ισχύει όμω, και άρα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την Εξεταστική Επιτροπή. Και άρα κατάλληλη επιτροπή είναι η συμβουλευτική, την οποία και προτείνουμε. Τέθηκε μια ερώτηση για τη νομική βάση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης Λισαβόνας. Όντως είχαμε μία νομική γνωμάτευση που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση αυτού του κανονισμού δεν είναι σωστή αυτή η νομική βάση, γι' αυτό συμφωνούμε με την κατάργηση. Η κατάργηση όμως της νομικής βάσης δεν αποκλεί τη δυνατότητα ο κανονισμός αυτός και χωρίς νομική βάση να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους δράσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούν ξαναζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Είχα πει ότι στο μέλλον αντιμετωπίζουμε μια τεράστια άξιο των θαλασσίων μεταφορών. Και μάλιστα σε δυσκολότερες περιοχές, είτε είναι ο Βόσπορος, είτε άλλες στενότερες θαλάσσιες οδούς. Η αλία λοιπόν όταν υπάρχουν θαλάσσια ατυχήματα ε, υποφέρει περισσότερο από, από όλους. Ε, ζημιώνεται το μέγι, περισσότερο από όλους τους άλλους. Γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να αυξήσουμε την ε, ε, θαλάσσια ασφάλεια στις μεταφορές. Αυτό βέβαια αφορά και την Επιτροπή Μεταφορών. Όταν έχουμε περισσότερες στενές, στενά περάσματα, θαλάσσια περάσματα, πρέπει να αυξάνεται η ασφάλεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ήθελα να απλώς να συμπεριλάβετε και αυτό το επιχείρημα. Συγγνώμη. Κανένας ε, δεν ε, ζήτησε να αποκλειστεί η Επιτροπή Μεταφορών, απλώς εκδικούμε και το δικό μας ρόλο. Δεν ε, θίξαμε εμείς την Επιτροπή Μεταφορών. Αυτοί ήθελαν να μας αποκλείσουν. Είναι δυνατόν να είμαι τόσο κοντόφθαλμη και να μην μπορώ να αναγνωρίσω το ρόλο των μεταφορών στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Αντίθετα, η Επιτροπή Μεταφορών είναι αυτή που δεν αναγνωρίζει το ρόλο της αλίας στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η κυρία η κυρία Δεν έχω να προσθέσω και πολλά. Σημείωσα προσεκτικά τα σχόλια των συναδέλφων. Σε ευχαριστώ θερμά όλους και ιδιαίτερα την υποστήριξη της διεκδίκησής μας ως συνδεδεμένης ε, επιτροπής με την Επιτροπή Μεταφορών. Είναι προφανές και υπάρχει αμέριστη υποστήριξη του θέματος αυτού ότι κατ' ουσίαν η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι κοινή και εγκάρσια και ο μοναδικός τρόπος να σεβαστούμε αυτή την εγκάρσια φύση της είναι να την αντιμετωπίσουμε ως τέτοια. Αν η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική εξεταζόταν μόνο από τη σκοπιά των μεταφορών, πραγματικά θα αλλοιωνόταν η ίδια η φύση της αυτή τη ε, θαλάσσια ολοκληρωμένη πολιτική. Μια και είναι ολοκληρωμένη, εγκάρσια, σφαιρική, θα πρέπει σφαιρικά να αντιμετωπίζεται και όχι μόνο υπό το πρίσμα των μεταφορών. Συμφωνούμε λοιπόν για αυτό το σφαιρικό χαρακτήρα. Η θέση τη επιτροπή Μεταφορών ε, δεν μα βρίσκει σύμφωνο και η διάσκεψη των Προέδρων, είπαμε, ανέβαλε την απόφασή τη. Εγώ δυστυχώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη για την έκβαση αυτή τη ε, αντιπαράθεσης. Και όχι μόνο για αυτόν τον κανονισμό, οι συνέπειες θα είναι σημαντικές για το σύνολο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Αν κάποια επιτροπή δικαιούται συμμετοχή εδώ, είναι η Επιτροπή Ελίας. Αλλά δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την ε, συνεργασία και τη να συνδεθούμε με την Επιτροπή Μεταφοράς. Και η απόφαση θα έχει συνέπειες όχι μόνο για την έκθεση και για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αλλά και για όλη την έκβαση των εργασιών μας και την προσπάθειά μας συνεργασίας με την Επιτροπή Μεταφορών ή με άλλες μεταφορές για αντίστοιχα θέματα που θα προκύψουν. Με άλλες επιτροπές, συγγνώμη. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως χαίρομαι που τουλάχιστον εμείς είμαστε σύσσωμοι υπέρ του αιτήματο της Επιτροπής Αλίας να γίνει συνδεδεμένη η Επιτροπή με τις μεταφορές για το θέμα αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω στους συναδέλφους και στην Επιτροπή είναι ότι επουδενή δεν θέλουμε κολλησιεργία ή να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι ε, πήγε αυτό το θέμα, γιατί στις 31 Δεκεμβρίου 2010 λύγει η χρηματοδότηση, οπότε σε καμία περίπτωση εμείς ε, δεν θα καθυστερήσουμε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τον κύριο Πένας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα επανέλθουμε στην έκθεση αυτή στην επόμενη μας συνεδρίαση, όπου θα δούμε και το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε αρκετά καθυστερημένοι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ, θέλω να επιταχύνουμε λίγο. Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, πρωτόκολλο με τις Αιχέλες. Δεν έχουμε ορίσει ακόμη εισηγητή. Το ΕΛΚ θα ορίσει εισηγητή για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας υποβάλει την πρότασή της για το νέο πρωτόκολλο με τις Ειχέλες. Ο κύριος Αλεξάνδρου έχει το λόγο. Oui, madame la présidente. C'est un accord. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία με, την, ε, με τις Ειχέλες. Ε, είναι η σημαντικότερη συμφωνία που έχει ποτέ συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα και αυτή η συμφωνία με τις αιχέλες είναι τμήμα του δικτύου των συμφωνιών ε, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο ε, στον Ειδικό Ωκεανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κοινοτικό στόλο, αλλά και για τις αιχέλες. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία του νέου αυτού πρωτοκόλου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο με τις αιχέλες. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο διάρκειας τριετούς. Ένα πρωτόκολλο που προβλέπει αλλιευτικές δυνατότητες για 48 ε, και 12 ε, παραγαδιάρικα. Ε, το, το ΝΑΖ όμως θα μειωθεί σε σχέση με, την, με το προηγούμενο πρωτόκολλο. Ε, το, το ΝΑΖ αναφοράς πέρασε πέρασε από 53.000 σε 52.000 τόνους ε, στο ε, νέο πρωτόκολλο και έγιναν διαπραγματεύσεις με τις Αιχέλες γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία μείωση των ε, αλλιευμάτων που εν μέρει οφειλόταν στον αρνητικό αντίκτυπο της πειρατείας στο τμήμα αυτό του Ινδικού ωκεανού. Ε, πειρατεία που βέβαια ε, πλήττει και τις ε, μεταφορές σε γενικές γραμμές αλλά και την ίδια την Αλλία Η χρηματική αντιπαροχή που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε βασιζόμενη στη διάκριση μεταξύ του του ε, υποστήριξη, της υποστήριξης του κλάδου είναι 5.600.000 ε, και ήθελα να πω ότι τα δικαιώματα πρόσβασης είναι 3.390.000 και η υποστήριξη του κλάδου είναι 2.220.000 ε, ευρώ σκοπό έχουμε να ενθαρρύνουμε την βιώσιμη και υπεύθυνη αλία στην περιοχή και είναι προφανές ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν για την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση μιας πολιτικής ε, ανάπτυξης ε, ε, της αλίας στις Αιχέλες, όμως είναι μια σημαντική συνεισφορά. Οι αλλιευτικές άδειες ε, δίδονται μετά από προκαταβολή που καταβάλουν ε, οι πλειοκτήτες. 61.000 ευρώ ανασκάφος αναέτος. που ε, υπολογίζεται βάσει ενός τονάζ αναφοράς. Δεδομένου λοιπόν του σημαντικού αυτού ποσού που είναι προκαταβολή και σας επισημαίνω ότι είναι προκαταβολή, για τα δικαιώματα πρόσβασης, εμείς ε, τελικά ε, καταλήξαμε να γίνουν δύο καταβολές. Για την πρώτη καταβολή δεν έχω ακριβώς αριθμητικά στοιχεία υπόψη μου, αλλά θα γίνει στην αρχή και η δεύτερη καταβολή θα γίνει μεσοπρόθεσμα Επίσης, ε, δύο ναυτικοί ε, από τις Σεϊχέλες ανασκάφος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να ενθαρρύνουμε μια αλλιευτική πολιτική αποτελεσματική και για τις για το, για το στόλο των Σεϊχελών, πρέπει βεβαίως να συνεισφέρουμε και στην κατάρτιση των ε, ναυτικών. Λοιπόν, δύο ναυτικοί ανασκάφος, δεδομένου τον αριθμό, του αριθμού των ε, αλλιευτικών σκαφών ε, που θα αλλιεύσουν στην περιοχή, ε, πρόκειται να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ο πληθυσμός των ζεϊχελών είναι αρκετά περιορισμένος και αν δεν κάνω λάθος, Πρόκειται για περίπου 80.000 άτομα. Βλέπετε λοιπόν τον αντίκτυπο, τον πραγματικό αντίκτυπο τέτοιου είδους μέτρων στην ε, οικονομία των Σεϊχελών. Επίσης προβλέψαμε στο πλαίσιο της πολιτική μας ε, στον Ινδικό ωκεανό να ενθαρρύνουμε το περιφερειακό πρόγραμμα εποπτείας, το οποίο συμμετέχουν οι τέσσερις χώρες με τις οποίες έχουμε αλληλευτικές συμφωνίες. Εμείς συνεισφέρουμε οικονομικά στο περιφερειακό πρόγραμμα εποπτείας ε, της Αλίας ε, και οι Σεϊχέλες, οι Μαδαγασκάρι οι Κομόρες ε, και συνεισέφεραν με το δικό τους τρόπο και έτσι μπορέσαμε στο πλαίσιο του περιφερειακού αυτού προγράμματος να αναπτύξουμε δράσεις αποτελεσματικές με αποτέλεσμα να πλήξουμε την παράνομη άναρχη και ελαφραία αλληλεία, δηλαδή ε, σκαφών που παρανόμως αλλιεύουν ε, ε, παραβιάζοντας όλες τις διατάξεις που αφορούν την αλληλεία στη ζώνη της Μαδαγασκάρης, των Σεϊχελών ή ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα. Κάναμε λοιπόν συγκεκριμένες αναφορές στις διατάξεις, της... Ε, IOTC, δηλαδή της Επιτροπής της Διεθνούς για τον Ινδικό Ωκεανό. Γνωρίζετε ότι η Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας για την περιοχή αυτή προβλέπει κάποιες, κάποιο, το κλείσιμο κάποιων αλλιευτικών ε, ζωνών, περιορισμένη δηλαδή αλία και όλα αυτά για να ε, ενθαρρυνθεί η υπεύθυνη αλία και τα ηχθίδια, ο πληθυσμό των ηχθιδίων. Ελπίζω ότι σας παρουσίασα επαρκώς το νέο αυτό πρωτόκολλο και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάντεξ. Ο κύριος κατέγ. Δεν ξέρω αν θα είμαι ενθουσιώδης, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Πρόκειται, όπω είπε και ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είναι για μια πολύ σημαντική συμφωνία και για μα αλλά και για, την, ε, για τι Αιχέλε, γιατί μιλάμε για 40 ε, γρηγροί και 12 παραγαδιάρικα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία ε, εκπροσωπούνται στο στόλο αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το πρωτόκολλο. Επίσης είναι και 63 εκατομμύρια τόνοι αλευμάτων ε, κα, και 5.350.000 ευρώ. Ένα τμήμα της κλιματικής αυτής αντιπαροχής ε, αποδίδεται στην τομεακή βοήθεια, κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ε, υπενθυμίσατε τον αριθμό των ναυτικών ανασκάφος, ε, δύο ναυτικοί από τις Αιχέλες ανασκάφους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πραγματικά ένας ε, πολιτισμός 80.000 ε, στις ε, Σεϊχέλες, αρκετά νέων, επομένω δύο ναυτικοί από τις Σεϊχέλες σε κάθε σκάφος είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Όσον αφορά τώρα την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία, δικαίως αναφέρατε την εποπτεία, Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε στην οργάνωση της ε, περιοχής, ε, όπως επίσης και στην προστασία των αλλιευτικών πόρων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική από οικονομικής απόψεως, αλλά και από κοινωνικής και από ανθρώπινης απόψεως ε, η συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά και για την αλληλεία των συγχελών. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε ορθά επί της συγκεκριμένη εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι δεν μακρηγόρησα. Ωραία, κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, η συμφωνία αυτή είναι η πιο σημαντική για την Ευρώπη, η πιο σημαντική για την Ισπανία και ιδιαίτερα για τα βασικά θυναλιευτικά, που είναι κυρίως ε, τα σκάφη που αλλιεύουν εκεί. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δεν πρόκειται να τα επαναλάβω. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το παράρτημα που υπάρχει για την πρόθεση της υπεύθυνη αλίας στα χωρικά ύδατα των Σεϊχελών και τη συμβολή μας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Γιατί όχι μόνο προχωρώνονται τα, τα σκάφη γρηγρή και παραγαδιάρικα να προσλαμβάνουν δύο ντόπιου ναυτικούς, αλλά συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη της συντήρησης των αλληλευτικών αποθεωμάτων και της ε, παιδεία αυτή υπέρ τη συντήρηση. Βέβαια, στον Ειδικό Ωκεανό είχαμε το ατυχές φαινόμενο της πειρατεία τον τελευταίο καιρό και έτσι δικαιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ο περιορισμός της χωρητικότητας του τονάζ. Θα ήθελα να επιμείνω στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ίσως και στο ψήφισμα που υιοθετήσαμε για την πειρατεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε τους ευρωβουλευτές ότι τα πλοία αυτά, και μάλιστα ένα από αυτά που είχαν απαχθεί από τους πειρατές, το βασικό σκάφος Αλακράνα, αλίευαν δυνάμει αλλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς θέμα αυτό. Μιλήσατε για κατάσχεση των παράνομων ε, σκαφών που αλίευαν χωρίς άδεια στα χωρικά αυτά ύδατα. Τι σημαία αυτά τα σκάφη. Ήταν ευρωπαϊκά τα σκάφη που αλίευαν παράνομα. παράνομα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε αύξηση ή μείωση του ποσοστού των παράνομων σκαφών μετά τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την Επιτροπή, προς την Κομισιόν. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τη συμφωνία, όσον αφορά την απασχόληση των, του πληθυσμού των ντόπιων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι προοπτικές ε, υπάρχουν για αυτό το θέμα της απασχόλησης του ντόπιου πληθυσμού. Και εγώ έχω κάποια σχόλια. Καταρχήν μια ερώτηση για τα παραγαδιάρικα. Αυξάνεται ο ρυθμό των παραγαδιάρικων. Ενώ η έκθεση αξιολόγησης, στη σύνοψη που έχουμε λάβει, αναφέρεται ότι η χρήση αυτών των δυνατοτήτων αλλιές από τα παραγαδιάρικα ήταν μικρό αναφέρω 262 τόνοι το 2007. Και υπήρξε μείωση των αλλιευμάτων εξαιτίας και της πειρατείας μεταξύ άλλων. Εξαιτίας της πειρατείας δεν εξαντλήθηκαν οι ελευτικές δυνατότητες, περιορίστηκαν και το 2000 είχαμε αύξηση από 52 σε 63.000 ε, ε, τόνους. Αλλά τελικά ούτε τους 63.000 τις ε, εξαντλήσαμε, γιατί παρόλο που τα γρηγροί είχαν 78% χρήση των αλληλευτικών δυνατοτήτων, τελευταία χρόνια υπήρξε μείωση αυτών των αλληλευτικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όχι μόνο για τον ευρωπαϊκό θυναλευτικό στόχο, αλλά και τη θετική, τις θετικές του συνέπειες στην τοπική βιομηχανία των Σιχελών. Γιατί ουσιαστικά η τοπική βιομηχανία χρησιμοποιεί το υλικό, τα, τα που, που εκφορτώνονται στη χώρα αυτή. Οπότε η έλλειφτη και αυτή η συμφωνία θα έχει άμεσο αντικτύπο και στο ΑΕΠ της χώρας αυτής. Γύρω στο 20% αναφέρεται, αλλά στην πράξη είναι πολύ νότερο αυτό το ποσοστό. Γιατί το λιμάνι ΜΑΕ ή το λιμάνι Βικτόρια που είναι ε, το σημαντικότερο λιμάνι της νήσου ΜΑΕ είναι το μοναδικό σημαντικό λιμάνι, το σημαντικότερο λιμάνι του Ινδικού. Στο λιμάνι αυτό της Βικτόρια συγκεντρώνεται όλος ο ευρωπαϊκός στόλος που αλλιεύει στα χωρικά ύδατα των Σιχελών, γιατί είναι το μόνο λιμάνι που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και μάλιστα η έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται σε 2.900 θέσει εργασίας που δημιουργούνται μόνο σε υπηρεσίες που παρέχονται σε ευρωπαϊκά σκάφη, αλλά και για την ε, μεταποίηση των αλληλευτικών προϊόντων. Οπότε η σημασία, οι συνέπειε δεν είναι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στις επίγειες δραστηριότητες, στον ανεφοδιασμό των σκαφών, στη μεταπητική βιομηχανία. Όλα αυτά δείχνουν το σημαντικό αντίκτυπο της Ελληνική αυτής συμφωνίας για την οικονομία των Σεϊχελών. Βέβαια, αναφέρθηκε το θέμα της πειρατείας και η πειρατεία μπορεί να απομακρύνει τον αλληλευτικό μας στόλο από εκεί, αλλά αυτό θα είναι πολύ αρνητικό όχι μόνο για τι Σεϊχέλε, αλλά για την ευρύτερη ζώνη. Και θα είναι πολύ σοβαρό ο αντίκτυπο μια πιθανή αποχώρηση του ελευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή. Γιατί ο ελευτικός μας στόλος συμβάλλει πέραν τη αναπτυξιακής βοήθεια που χορηγούμε. επίση ό,τι αφορά τι προκαταβολέ που οφείλουν να καταβάλουν ε, τα γρηγρή των 61.000 ευρώ. Το 50% αυτό που προβλέπεται είναι ένα πάγιο κατά αποκοπή Σας έχω σχεδόν απόλυτη εμπιστοσύνη κύριε Αλεξάνδρου γιατί σα γνωρίζουμε πολύ καλά. Ελπίζω, ελπίζω να τεθεί άπαξ και διαπαντός ε, τέρμα στην ε, αντιπαράθεση που υπάρχει με την κυβέρνηση των Σεϊχελών για τα λιεύματα. Γιατί από 21.000 που ήταν αρχικά ε, φτάσαμε σε 61.000. Τριπλασιάστηκε αυτό το ποσό. Ελπίζω, ελπίζω, αν γίνει δεκτό τελικά αυτό το μέτρο, να σταματήσουν πια οι διεξυπισμοί που είχαμε με τις Ειχέλες ε, για τις δηλώσεις. Μου λέτε ναι, σας έχω εμπιστοσύνη και ελπίζω ότι έτσι έχει λύθει το πρόβλημα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Κύριε Αλεξάνδρου, έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ξεκινήσω με το τελευταίο σας ερώτημα. Να σας καθησυχάσω. Το νέο ποσό των προκαταβολών που είναι 61.000 ευρώ είναι η ολοκλήρωση της συζήτησης και της διαμάχης που είχαμε, που είχαμε εδώ και δύο χρόνια με τις αρχές των Σεχελών για τις προκαταβολές. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και το οποίο ανταποκρίνεται στο, στα, στα μέσα, στο, στο μέσο όρο των αλλιευμάτων ε, του κοινοτικού στόλου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον κανένας προβληματισμός, καμία διαμάχη. Βέβαια αυτό δεν ότι στο μέλλον ενδεχομένως. Ε, οι αρχές των Χελών θα έρθουν μία μέρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με νέα αιτήματα. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό που έγινε στο πλαίσιο των προκαταβολών με τις Σεϊχέλες αποτελεί μία πρόοδο πολύ σημαντική και γνωρίζουμε ποιο είναι το κόστος του ευρωπαϊκού ε, στόλου, αλλά θελήσαμε με την καλή έννοια να παίξουμε με τις αρχές των Σεϊχελών και καταλέξαμε σε αυτό το ποσό, μιλάω για, τις 61, για τα 61.000 ευρώ, που δεν ε, το αποφασίσαμε το Μάιο, αλλά ήταν αντικείμενο ιδιαίτερη συνεδρίαση της Επιτροπής της Μικτή ε, το Δεκέμβριο του 2009, μια συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν οι ε, εκπρόσωποι των χωρών μελών που συμμετέχουν ε, στην Αλία στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Όσον αφορά τώρα τον αντίκτυπο στον τομέα της απασχόλησης, μίλησα για το ε, θέμα ε, της, των ναυτικών στο πλοίο, εν πλώ. Υπάρχει λοιπόν ένας αντίκτυπος σφαιρικότερος βέβαια ε, στην τοπική δραστηριότητα των Σεϊχελών και λόγω του λιμανιού του ΜΑΕ ε, όλα τα θυναλιευτικά, όλα τα θυναλιευτικά που ε, ε, αλλιεύουν στην περιοχή κάνουν μία στάση στο ΜΑΕ είτε για να αλλάξουν πλήρωμα είτε για ανηφοδιασμό και εκατοντάδες, δεν έχω ακριβώς βέβαια τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, πάνω από χίλια άτομα ε, εργάζονται και γνωρίζετε ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτές τις χώρες ενός μισθού. Ένας μισθός μπορεί να ε, θρέψει πολλά μέλη μιας οικογένειας. Και αυτό το λέω και για τον ανεφοδιασμό των σκαφών. Υπάρχει επίσης η αλλαγή του προσωπικού, ο ε, ο ανεφοδιασμός ε, εν πλώ και λοιπά. Ε, όπως είπατε και εσείς, ο αρνητικός αντίκτυπος της πειρατείας έχει οπωσδήποτε αρνητικές συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο για τις Σεϊχέλες. Και οι Σεϊχέλες ήταν η πρώτη χώρα της περιοχής που επλήγει από την... από τη μάστιγα της πειρατείας. Αλλά το είπα και στην παρουσίασή μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε εκτός από τη συμφωνία, ε, την αλληλευτική συμφωνία και ένα πρόγραμμα περιφερειακό εποπτείας που καλύπτει όλη την περιοχή, τη δυτική του Ινδικού ωκεανού με σκοπό να αποθαρρυνθούν ε, οι δραστηριότητες παράνομης λαθιαία και Άναρχη αλληλεία. Ε, δεν υπήρξαν ευρωπαϊκά σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία ε, που να προέβησαν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Υπήρξαν όμως πάρα πολλά σκάφη ε, τρίτων χωρών ε, που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, όπως επίσης και προέβησαν σε παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις σας. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη μας συνεδρίαση. Περνάμε στο σημείο 8 τώρα το νέο πρωτόκολλο για τις αλληλευτικές ε, δυνατότητες και την χρηματοοικονομική σύμβολη με την ε, δημοκρατία του Σαντομέ και Πρίσιπε. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Καπόλα Σάντος. Θα είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ε, τριετές πρωτόκολλο που συνεχίζει το προηγούμενο πρωτόκολλο του 2006, για το οποίο ήμουν και πάλι συγκεκριτής εγώ. Το πρωτόκολλο προβλέπει δυνατότητες ελευτικές σε 40 ελευτικά σκάφη, τρία λιγότερα δηλαδή από ό,τι στο προηγούμενο, με ε, χωρητικότητα αναφορά σε 70.000 τόνους. Η χρηματική αντιπαροχή θα είναι λίγο υψηλότερη από την προηγούμενη, με ποσοστό γύρω στο 40%, με στόχο την ανάπτυξη του ελευτικού κλάδου, λίγο λιγότερο δηλαδή από το προηγούμενο πρωτόκολλο και θα Ήθελα να δούμε γιατί. 35 ευρώ τον τόνο είναι η συμβολή των πλειοκτητών και θα ήθελα να σας επισημάνω το εξής. Συζητούμε αυτή την έκθεση χωρίς να έχουμε λάβει μέχρι στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οποιαδήποτε επίσημη αναθεώρηση της απόφασης του Συμβουλίου. Επίσης δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως πληροφορία ούτε για αξιολόγηση, ούτε καμία άλλη ενημέρωση. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα θέσουμε το απόγευμα στην Επίτροπο Δαμανάκη. Γιατί πραγματικά είμαστε δυσαρεστημένοι από αυτή την έλλειψη ενημέρωσης που δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτά κυρία Πρόεδρε και περιμένουμε την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποια σχόλια όμως και θα ήθελα απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ ότι ούτε καν τη σύνοψη για την εξπόστα αξιολόγηση δεν λάβαμε για το Σάντο Μέι Πρίσιπε. Ενώ για τις Αιχέλες λάβαμε μια τέτοια σύνοψη. Έχουμε μόνο την ενημέρωση για μια συνεδρίαση τη Μικτή Επιτροπής. Έχουμε ελάχιστη ενημέρωση. Πώς θα κάνουμε την αξιολόγηση αυτού του πρωτοκόλου. Επιπλέον έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ήταν τόσο χαμηλή χρησιμοποίηση όσο αφορά τη συμφωνία αυτή από τη Μικτή Επιτροπή. Γύρω στο 10% αναφέρεται το ποσοστό χρησιμοποίησης. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό το στοιχείο, αλλά εγώ αυτό έμαθα. Είναι σωστή αυτή η πληροφορία. Επίσης, γιατί αυτό το χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της συμφωνίας, όταν γενικώ υπάρχει Έτοιμα διόν από τον Ατλαντικό για να πάνε στον Ειδικό εξαιτία της, ε, της πειρατείας. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει αυτή η χαμηλή εφαρμογή της συμφωνίας, η χαμηλή χρήση. Η Μικτή Επιτροπή αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που ανέκυψε με το σύστημα UBMS. Λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί μας είχαν πει τότε ότι δεν λειτουργούσε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να διευκολύνει την κυβέρνηση του Σαν και Πρίνσιπε, προκειμένου να δοθούν ενισχύσεις για να λειτουργήσει το σύστημα UBMS. Τελικά τι έγινε, άρχισε να λειτουργεί ή έμεινε α, δυσλειτουργικό. Υπό αυτέ τι συνθήκε είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε την αλληλευτική συμφωνία, γιατί δεν υπήρξε σχεδόν ενημέρωση. Αλλά αυτό θα το θίξουμε το απόγευμα στην αρμόδια επίτροπο δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση ότι φορά τι διεθνεί ελευθερικέ συμφωνίε. Κύριε Αλεξάνδρου, έχετε το λόγο. Oui, madame. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για τη μη παρουσίαση από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέσεις αξιολόγησης. Γνωρίζετε ποιοι είναι οι λόγοι. Περιμέναμε τη συμφωνία, τη διοργανική, σε σχέση με την ε, ε, υποβολή των ε, και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι δεν λάβατε εγκαίρως τα έγγραφα αυτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ε, στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι μία συμβιβαστική λύση θα ε, βρέθηκε και ότι ε, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να σας υποβάλουμε τα συγκεκριμένα έγγραφα. Δεν πρόκειται για μπλοκάρισμα ούτε από δική μου πλευράς, ούτε από πλευράς υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα ε, θέμα που έχει, που έχει να κάνει με ε, μια πολιτική, ένα ευρύτερο θέμα, εν πάση περιπτώσει, πολύ πέρα από τις αλληλευτικές συμφωνίες. Αλλά καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας λόγω του ότι δεν λάβατε αυτές τις ε, ex post ε, εκθέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αξιολογήσετε αντικειμενικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων πρωτοκόλων. Τώρα για τα ερωτήματα της μείωσης της ε, χωρητικότητας αναφοράς. Πέρασε από 8.500 τόνους σε 7.000 τόνους το νέο πρωτόκολλο και ο βασικός λόγος είναι ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ λίγο και τα σκάφη έπαιρναν άδειε, αλλά τελικά δεν αλλίευαν υποχρεωτικά ε, στην ε, ε, ζώνη την αλλιευτική του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Δυστυχώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναθεωρήσουμε προς τα κάτω τον αριθμό ε, το, τη χωρητικότητα αναφοράς και δεν σας κρύβω την αρχική πρόθεση που ήταν ε, να έχουμε μια χωρητικότητα αναφοράς που θα ήταν ακόμη χαμηλότερη από τους 7.000 τόνους. Αλλά γνωρίζετε ότι για τις διαπραγματεύσεις χρειάζονται δύο μέρη και αυτός ο αριθμός 7.000 τόνοι ε, αντιστοιχεί στο μέγιστο που μπόρεσε να παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελάχιστο που μπόρεσαν να δεχθούν ε, οι αρχές του ΣΑΟΤΟΜΕ και Πρίνσιπε στις διαπραγματεύσεις. Όμως αυτό θα ε, δώσει τη δυνατότητα μια, μιας περαιτέρω ε, αποστολή σκαφών ε, αν η κρίση της πειρατείας συνεχίσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδιπλωθούμε ε, προοδευτικά ε, στην περιοχή του Ινδικού ωκεανού. Όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, πρέπει να σας πω το εξής, ότι το προηγούμενο πρωτόκολλο είχε προθεσμία 31 Μαΐου 2010 και περιμέναμε το Φεβρουάριο ρωτήσαμε τις αρχές, ε, ζητήσαμε από τις αρχές του Σάουτο και Πρίνσιπε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να έχουμε ένα νέο πρωτόκολλο την στιγμή της εκπνοής του προηγούμενου πρωτοκόλλου. Αυτό ήταν αδύνατον γιατί οι αρχές του ΣΑΟΤΟΜΕ με και Πρίνσιπε ε, ισχυρίστηκαν ε, λόγους χρονοδιαγράμματος και δυστυχώς αυτό καθυστέρησε την ε, ε, μονογραφή του πρωτοκόλου που έγινε τελικά 15 Ιουλίου 2010, δηλαδή σχεδόν δύο μήνες μετά από την ε, λήξη του προηγούμενου πρωτοκόλου. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει ένα νομικό κοινό που βάσει της ρήτρα αποκλειστικότητας παρεμποδίζει τα σκάφη να αλλιεύσουν με ιδιωτικέ άδειες όσο η διαδικασία ε, για την ε, προσωρινή διαδικασία και για τη σύναψη του πρωτοκόλλου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή ήταν ε, μία πληροφορία που έπρεπε να σας δώσω για να προκαταβάλω, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσατε να είχατε θέσει. Σε σχέση με τις διάφορες ερωτήσεις, αυτά είχα να πω. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ευχαρίστω να απαντήσω. Thank κύριος Αρσένης. Ευχαριστώ. Για το ίδιο θέμα και πάλι. Σε ήθελα να αναφερθώ στην έλλειψη της αξιολόγησης, της έκθεσης αξιολόγησης. Ίσως υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που δεν την έχουμε στα χέρια μας. Uh, θα ήθελα όμως να έχουμε την έκθεση αξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και κλείνει το μικρόφωνο. Α, ε, χωρίς αυτή την έκθεση αξιολόγησης δεν μπορούμε να, έχουμε, να κάνουμε σωστή δουλειά. Το είπα κύριε Αρσένη. Ο κύριος Αλεξάνδρου είναι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα λάβει θέση. Είπε ότι καταλαβαίνει ότι χρειαζόμαστε την ενημέρωση αυτή, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Αυτό όμως θα το θίξουμε το απόγευμα στην αρμόδια επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη. Γιατί εκείνη θα πρέπει να δεσμευθεί απέναντί μας και εμείς απέναντί της. Άλλωστε, το είχαμε αναφέρει τις προάλλες με τους συντονιστές. Και θα προτείνουμε κάποιες αναλεκτικές λύσεις την κυρία Δαμανάκη το απόγευμα. Τι να μας πει ο κύριος Αλεξάνδρου. Δεν μπορεί να ταχθεί ούτε υπέρ ούτε κατά. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Σε άλλε αλληλευτικέ συμφωνίε είχαμε τουλάχιστον τη σύνοψη τη εξπόστη αξιολόγηση. Εδώ ούτε καν τη σύνοψη. Εν πάση περιπτώσει, σημείο 9 τη ημερία τη διάταξη. Συμφωνία για μέτρα του λιμένοντος, του προκειμένου να προληφθεί, αποτραπεί ή καταργηθεί παράνομη, λαθρέα και άναρχη ελεία. η καταργηθει παρανομη λαθρεα και αναρχη αιλια η επίτροπος, η συγγνώμη, πρόεδρος Επιτροπής είχε αναλάβει αυτό το θέμα. Η ΦΑΟ ενέκρινε το 2005 ένα σύστημα ε, μέτρων για ε, τον ε, λιμένα προκειμένου να παταχθεί η παράνομη λαθρέα και άναρχη αιλία. Προτινόταν μια ελάχιστη δέσμη μέτρων προαιρετικών και προτείνονταν η εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη. Το 2005 ήταν προαιρετικός αυτός ο μηχανισμός. Στη συνέχεια προτάθηκε ένα διεθνές ε, δεσμευτικό εργαλείο και έτσι το 2007 ελήφθη η απόφαση θέσπης αυτού του διεθνούς μέσου που θα είναι νομικός δεσμευτικό. Ήταν αρκετά χρονοβόρα η διαδικασία. Το 2008 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε μια απόφαση την οποία ε, την, ε, εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσει ε, για τη συγκέντρωση πληροφοριών για το έγγραφο αυτό, το οποίο υπεγράφει στη Ρώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευση Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το 2009 και θέλουμε να εγκρίνουμε οριστικά αυτή τη συμφωνία. Τα μέτρα για το λιμένα είναι πολύ σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μάχη ώστε στις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας να προταθεί αυτό το θέμα ως υποχρεωτικό και θα ήθελα ως συγγήτρια να υποβάλω μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διάβασα το έγγραφο της ΦΑΟ που θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ρώμης, στην οποία θα συμμετέχει εκ μέρους μας η κυρία Λόβιν. Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το έγγραφο της ΦΑΟ ότι υπάρχει εμφανής αντίδραση και αντίσταση ως προς τα μέτρα αυτά για το λιμένα εκ μέρους ορισμένων χωρών και αναφέρονται οι χώρες του ειρηνικού. Σας το είπα τις προάλλες και εγώ για την Παππούα Νέα Και στην Επιτροπή Κεντροδυτικού ε, Ειρηνικού υπήρξε κάθετη αντίδραση και αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, γιατί προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα συμβαλόμενα μέρη ως προς την εφαρμογή αυτών των μέτρων λιμένα. Αλλά οι χώρες Λατινικής Αμερικής αναφέρεται συγκεκριμένα η Αργεντινή αλλά γενικώ γίνεται λόγο για τη Λατινική Αμερική. Ποιε χώρε τη Λατινική Αμερική περιλαμβάνονται. Η Χιλή είναι από τι χώρε που ε, δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα λιμένα. Το λόγο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Νικολόβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την ε, επίσημη υπογραφή της συμφωνίας έχουμε τη Χιλή που έχει υπογράψει και το Περού η Ουργουάη από τις λατινοαμερικανικές χώρες. Καμία χώρα από τον Ειρηνικό, με εξαίρεση της νήσου Σαμόα και από τις αφρικανικές χώρες που είναι εταίροι μας, η Μοζαμβίκη έχει υπογράψει και οι παραδοσιακοί εταίροι μας, η Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Νέα Ζηλανδία και Ρωσία. Βεβαίω, η υπογραφή δεν σημαίνει και αυτόματη επικύρωση. Είναι όμως ήδη ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Μέχρι τώρα έχουμε 23 χώρες συνολικά που έχουν υπογράψει, δύο έχουν ενταχθεί και έχουμε ήδη 25 χώρες. Εάν και 25 επικυρώσουν, σημαίνει ότι η συμφωνία θα τεθεί ενισχύει. Ελπίζω να σας απάντησα. Όσον αφορά τώρα τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας, ξέρω ότι και εσείς και άλλα μέλη της Επιτροπής έχουν συμμετάσχει. Η επίσημη αποστολή ε, μέσα στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών συμφωνιών είναι να υιοθετήσει μέτρα για τις ε, χώρες αυτές και μέσα στα πλαίσια του IOTC δεν έχουμε επιτύχει ικανοποιητικά να υιοθετήσουμε τέτοια μέτρα μέσα στο πλαίσιο των άλλων συμφωνιών IATTC, διότι αυτές οι χώρες δεν έχουν ακόμα υπογράψει. Δεν έχουν ακόμα λοιπόν αποφασίσει αν είναι σωστό να συμφωνήσουν ε, ή όχι, να υπογράψουν ή όχι. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσουμε και να εξηγήσουμε καλύτερα αυτή τη συμφωνία μέσα στο πλαίσιο των περιφερειακών συμφωνιών αλίας για να πείσουμε τις χώρες αυτές ε, περιφερειακών οργανισμών αλίας για να μπορέσουν και οι χώρες αυτές να ενταχθούν και να επιτύχουμε τη συνολική επικύρωση της συμφωνίας όλων αυτών των χωρών. 25. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του κανονισμού του 2005 για την πάταξη της άνοχης παράνομης και ελαθρέας αλίας έχει κάποια μέσα εις βάρος των χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα αυτά. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η αλία που προέρχεται από τις χώρες αυτές είναι αλία που δεν εμπίπτει στην παράνομη λαθρέα και αναρχαιλία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα να εξαναγκάσει κατά κάποιο τρόπο ή να πιέσει τις χώρες αυτές να δεχτούν αυτά τα μέτρα. Αλλιώ θα μπορούσαμε να συντάξουμε ακόμη και κατάλογο μαύρη λίστα χωρών που δεν μπορούν να εξαγάγουν, να εξαγάγουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα τους βοηθήσουμε πραγματικά να καταπολεμήσουν την παράνομη αλληλεία και να έχουμε μία εξασφάλιση ότι τα ληφτικά αυτά προϊόντα δεν είναι προϊόντα παράνομης, λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Ευχαριστούμε κυρία Νικολόβα. Κύριε Αλεξάνδρου, μα έχουν απομείνει πέντε λεπτά. Δεν θέλω να υπερβούμε το ωράριο των διερμηνέων. Έχετε λοιπόν πέντε λεπτά για να μας μιλήσετε αν θέλετε για τη Βενεζουέλα. Την πρόσβαση λευτικών σκαφών με σημαία Βενεζουέλας. Μάλλον εύκολο είναι θέμα, πανεύκολο θα έλεγα. Έχετε ένα πεντάλεπτο και μπορείτε να μας κάνετε την παρουσίαση. Oui, ναι, κυρία Πρόεδρε, απλώ ενημερωτικά πρόκειται για την πρόσβαση από αλληλευτικά σκάφη της Βενεζουέλας ε, στις ακτές της Γουιάνας. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο για πολλά χρόνια είχε επιληθεί μέσω του κανονισμού ΤΑΚ και ποσοστώσεων. Μα έδινε τη δυνατότητα να δώσουμε άδειε αλίευση ε, στα σκάφη της Βενεζουέλα που αλίευαν στα ανοιχτά της ε, γαλλικής Γουιάνας παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε νομική συμφωνία μεταξύ ε, της ε, Βενεζουέλας και τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τότε που έγινε η συζήτηση για τα ΤΑΚ το Δεκέμβριο του 2009 αποφασίστηκε ότι έπρεπε να αλλάξει η κατάσταση και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια νομική βάση που να δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν ε, τα σκάφη της Βενεζουέλας ε, και να αλλιεύουν και να εκφορτώνουν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικός ο αντίκτυπος της αλλιευτικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων σκαφών της Βενεζουέλας σε επίπεδο εκφορτώσεων για, τις, ε, για τα εργοστάσια μεταποίησης. Ε, οπότε έπρεπε να διατηρηθούν οι δραστηριότητες αυτές. Και μετά από προβληματισμό μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε αυτή την έλλειψη νομικής συμφωνίας, χωρίς να γίνει όμως υποχρεωτικά μια συμφωνία αλλιευτική με την Γουιάννα. Ήταν λοιπόν δυνατόν να λάβει μία απόφαση το Συμβούλιο υπομορφή δήλωσης για την πρόσβαση των σκαφών της Βενεζουέλας στις ακτές της Γουιάνας. Αυτό θα, θα έδινε τη δυνατότητα να ε, μην έχουμε τη δυσκολία της νομικής συμφωνίας. Το ζήτημα εξετάζεται τώρα σε επίπεδο ε, νομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι θα είναι θετική η έκβαση Τη ανταλλαγή αυτή απόψεων και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Bueno, pues, eh, nada. ευχαριστούμε πολύ κύριε Αλεξάνδρου. Στην επόμενη συνεδρίαση ελπίζω να έχει ορίσει το αλκησηγητή για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ θερμά σε όλους. Η συνεδρία συλλύεται μέχρι τις 3. Παρακαλώ να είστε συνεπείς στο ραντεβού, γιατί θα έρθει η Επίτροπος Δαμανάκη.